Please take your... Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Wir haben Tagesordnungspunkt Nummer 1, Annahme der Σημείο 1 έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Η κυρία Σάκε λόγω άλλου κολλήματο δεν θα μπορεί να είναι παρούσα. Ε, το υπόλοιπο απόγευμα θα ήθελε να ψηφίσουμε αμέσως τη δική της έκθεση αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχω καμία απολύτως ανακοίνωση, οπότε μπορούμε να περάσουμε αμέσως στις ψηφοφορίες και περνάμε στο σημείο 6 που είναι η έκθεση της κυρίας Σάκε για την στρατηγική ψηφιακής ελευθερίας. Θέλετε να πείτε κάτι κυρία Σάκε. Πρώτου ληφθεί η οριστική απόφαση για έκθεσή σα. Δεν βλέπω να θέλετε. Ωραία. Ψηφίζουμε επομένω. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Γίνεται δεκτή. Τρεις υπέρ, δύο κατά, λέει ο πρώτος. Συμβιβαστική 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές έλεγχος ηλεκτρονικός πέρας προφορίες, 25 υπέρ 32 κατά απορρίπτεται. Προφορική 2 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 32 μόνο το δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην 33. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. 33. Λοιπόν, αρχίζει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 34-23 εγκρίνεται. 34 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Συμβαστική 4 υπέρ. Δεύτερο τμήμα της 34 ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας. 32 προς 24 γίνεται δεκτή. Γίνεται δεκτό το δεύτερο μέρος συγκεκριμένα. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι γίνεται δεκτή, αλλά θα κάνουμε έλεγχο. Πέρας. Δεν γίνεται δεκτή. 28-31. Απορρίπτεται. 39. 39, συγγνώμη. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στην... Όχι. Στην 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η 51 εκπίπτει, 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην 57 ψήφι υπέρ ψήφι κατά, αποχές απορρίπτεται. 58 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 60 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά αποχές έλεγχος. πέρας ψηφοφορίας. 37-25 γίνεται δεκτή. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. περας προφορια προφορίας ελέγχου. 29-24 γίνεται δεκτή. 8 βουλευτές δεν ψήφισαν. 64 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 66 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εδώ άλλαξε, άλλαξε τελείως το, το σύστημα. Θέλετε έλεγχο στην 67. Ωραία, άρχεται η ψηφοφορία. Η 68 έχει γίνει δεκτή. Πέρας. Δεκτή. 69 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Θα κάνουμε έλεγχο. 71. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 74 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 77 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 79 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 84 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά διαφορετικό το 87 θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά πέρας Απορρίπτεται. 31-32. Κύριε Σαλαφρανκά. Θα ήθελα να σας πω ότι τώρα έρχεται η κάρτα μου και εγώ ψήφισα, δεν καταψήφισα, απλώς θέλω να το λάβετε υπόψη μέχρι να έρθει η κάρτα μου. Καταψηφίζω λοιπόν. Ούτως ή άλλως είχε απορριφθεί. Τώρα απερίφθη με 31 υπέρ 33 κατά. Εγώ δεν ψήφισα. Όχι, είναι δικό σας πρόβλημα. Δεν δούλεψε το μαραφέτη μου. 32-33 τότε. dafür. 88 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 50, 95 ε, συγγνώμη. Εκπίπτει και αυτή. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Όχι, όχι. 102 είναι η επόμενη ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 105 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 106 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 108 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 110 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 112 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 113 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. 114 σε δύο τμήματα. Τμήμα 1. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Διπλό Πλήγμα για την τροπολογία λέει ο πρόεδρος. 115. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 116. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 117 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά από έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 32-31 γίνεται δεκτή. Κύριε Σαλαφράγκα. Όχι. 32-32 απορρίπτεται επομένω. επομένως. Σαλαφράγκα καταψήφισε. 10. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 11. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15. Υπέρ. 14 λέει πάλι ο πρόεδρος. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεκατέσσερα, ηλεκτρονικός έλεγχος, υπενθυμίζει ο πρόεδρος. Πέρας. Εγκρίνεται, 36-23. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Έχουμε τη γνωμοδότηση της ίντα τώρα. Ίντα 1, ψηφιπέρ, κατά αποχές δεκτή. 53 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τα 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, είναι τα 12 σε δύο τμήματα, πρώτο τμήμα, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε, το δεύτερο μονάχα, ψήφι υπέρ του δεύτερου τμήματος, κατά αποχές δεκτό, είναι τα 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας. Και ο κύριος Σαλαφράγκα υποστηρίζει 57 υπέρ, καμία ψήφος κατά και 5 αποχές. Συγχαρητήρια. Μπορείτε να πάτε λοιπόν στην επόμενη σας συνεδρίαση. Και ερχόμαστε πίσω στο σημείο 3, που είναι η έκθεση Ρουίτε Βάρισ. Θέλετε να λάβετε το λόγο σχετικά. Όχι. Ψήφισμα τότε. Παρακαλώ. 36 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικά, έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 48-8 δεκτή. ΔΕΒΕ 1. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά έλεγχος για τις 45 45 Ja, ist geschlossen. Πέρας προφορίας. 27 με 36 απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Με την ίδια πλειοψηφία. ...48. Η 47 είναι γλωσσικού χαρακτήρα, μονάχα μόνο για το γαλλικό κείμενο. ...48 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτη DB2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. DB3 υπέρ. Κύριε Ταβάρη, παρακαλώ. Από τη συζήτηση που είχαμε χτες, στην Επιτροπή Νομικών Επιθέσεων ε, για όλες ε, τις ε, τροπολογίες ΔΕΒΕ. Έχω την εντύπωση ότι κανένας, καμία ομάδα δεν έχει αντιρρήσει. Έτσι λοιπόν θα πρότεινα να τις ψηφίσουμε όλες σε ομάδα αν δεν υπάρχει αντίρρηση από τις πολιτικές ομάδες για να γλιτώσουμε χρόνο. Ισχύει αυτό για όλες τις τροπολογίες ΔΕΒΕ ή μόνο για αυτές που βρίσκονται εδώ. Μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις τροπολογίες της ΔΕΒΕ unblock. Ψήφι υπέρ. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις ε, για τις τροπολογίες της ΔΕΒΕ. Δεν ισχύει. Λοιπόν, ας ψηφίσουμε σε μπλοκ. Λοιπόν, ΔΕΒΕ 2 έως ΔΕΒΕ... 2 ΔΕΒΕ 12. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. <laughs> Για την 4 υπήρχαν πολλέ ψήφοι κατά, αλλά καταφέραμε να έχουμε πλειοψηφία, λέει ο κύριο Μπροκ. Ψηφίσουμε για την 4 χωριστά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική 1 υπέρ. Μάλιστα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η σχεδίση εισηγητρία της ομάδας μου αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε άλλη ψηφοφορία στην Επιτροπή Ελευθεριών και είναι κατά τη παρουσίαση αυτή τη ψηφοφορική τροπολογία και το ίδιο ισχύει και για την προφορική τροπολογία περιθμών 2. Ευχαριστώ. Κύριε Σταβάρες, ε, ναι, πρόεδρε. Είχαμε μια συνάντηση με την ε, σκιώδη συγκεκριά του ΕΛΚ και η συνάδελφος Κίνγκα Γκάρντ και μας είπαν ότι θα καταψήφιζε το ΕΛΚ την τροπολογία αλλά όχι κατά της παρουσίασης της τροπολογίας. Έτσι λοιπόν, ε, εγώ δέχτηκα τις προφορικές τροπολογίες του ΕΛΚΟ συγητής ε, από τεχνική σκοπιά. Νομίζω ότι θα πρέπει να ψηφίσει κάθε ομάδα ανάλογα με τη γραμμή τη όλε αυτέ τι τροπολογίε. Αλλά θέλω να τονίσω το εξή. Αυτέ οι τρει τροπολογίε αφορούν του πρόσφυγε. Ε, και θα ήθελα να πω ότι δεν εννοούμε μια διευρυμένη έννοια του πρόσφυγα, αλλά μιλάμε εδώ για έναν ορισμό αρκετά περιορισμένο. Αναφερόμαστε σε ανθρώπου που έχουν κάρτα, που έχουν ταυτότητα από την είπατε του ΙΕ για τους πρόσφυγες. Επομένως μιλάμε για μια ερμηνεία πολύ περιορισμένη. Ο κύριος Σαλαφράγκα. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την αντίρρησή μου γενική φύσεως ε, στο να φέρνουν αντίρρηση οι ομάδες στην παρουσίαση προφορικών τροπολογιών. Μίλησα όμως εγώ με τη σκοντή συγγήτρια και είναι αντίθετη βέβαια. Ε, ξέρουμε σε σχέση με την τροπολογία 13 ότι θα τη χάσουμε, αλλά αυτές τις πληροφορίες έχω λάβει εγώ από τη δική μου ομάδα. Επομένως, η δική μου ομάδα είναι κατά τροπολογιών 1 και 2. Συγγνώμη, Πρόεδρε, λέει ο κ. Σταβάρες. Σέβομαι τις πληροφορίες ε, που μας δίνει ο κύριος Ελαφράνκα, αλλά εμείς δεν λάβαμε τέτοια ενημέρωση σήμερα το πρωί. Ε, υπήρξε ένα συμβασμό και εγώ δέχομαι ως ηγητής της τροπολογίας του ΕΛΚ και θα ήθελα να έχω ενημέρωση από τη γραμματεία αν μια πολιτική ομάδα μπορεί να φέρει αντίρρηση μιας για να παρουσιαστεί ε, μια προφορική τροπολογία από έναν εισηγητή. Από όσο γνωρίζω, ο εισηγητή είναι αυτό που μπορεί να φέρει αντίρρηση στην κατάθεση προφορικών τροπολογιών από μονομένα μέλη και στην Ολομέλεια χρειάζεστε 40 βουλευτέ. Αλλά θα ήθελα να μου απαντήσει η γραμματεία. Συγγνώμη, πρέπει να υπενθυμίσω του κανονισμού. Δεν ξέρω τι έχει γίνει μεταξύ σκιωδών εισηγητών και τι συμφωνίες έχουν ε, υπάρξει. Ο κανόνας είναι σαφής ότι εάν υπάρξει αντίδραση μιας ομάδας, τότε δεν μπορεί να ψηφιστεί η τροπολογία. Και για μένα έχει τελειώσει το θέμα επομένω. Μπορείτε να την καταθέσετε και πάλι στην ε, Ολομέλη αυτή την τροπολογία. Ο κύριος Σταβάρες, ε, θέλω μια διευκρινήση ότι πράγματι αυτό λέει ο κανόνας. τότε να γραφεί στα πρακτικά ότι πρόκειται εδώ για αντιστροφή ενός συμβιβασμού, ο οποίος επιτεύχθη μόλις ε, πριν μια-δυο ώρες, χωρίς καμία ενημέρωση του συγκητή. Ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι σαφής, δεν καταγράφονται οι συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί η οποιαδήποτε πολιτική ομάδα να αλλάξει την άποψή της κατά Μπορεί να δεχτεί μια συμφωνία, μπορεί να μην την ε, ε, δεχτεί, μπορεί να είναι καλό ή μπορεί να είναι κακό, ηθικό ή μη, αλλά ο κανονισμός δεν αναφέρεται στο θέμα αυτό. Όσο υπάρχει αντίρρηση μιας πολιτικής ομάδας, τότε δεν μπορούν να ψηφιστούν. Μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά είναι ένας προστατευτικός μηχανισμός κατά των ε, προφορικών τροπολογιών. Ψηφίζουμε την 52. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 53 εκπίπτει. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές δεν ήταν σαφές νομίζω ότι εγκρίνεται όμως ε? κύριε Σαλαφράγκα εγκρίνεται εντάξει καλά κάνουμε έλεγχο 58 έλεγχος περισσότερες ψηφοφορίας. ...31 ψήφοι υπέρ, 32 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά αποχές 59 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 60 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Σας παρακαλώ να σηκώνετε ψηλά τα χέρια σας όταν γίνεται η ψηφοφορία για να βλέπω. Ελπίζω ότι θα με βοηθήσετε όλοι με το να ψηφίσετε, γιατί δεν μπορώ να εκτιμώ τι θέλουν αυτοί που δεν σηκώνουν το χέρι τους. Πέρας. Εγκρίνεται 33-21. Όταν τρεις φορές ζητήσει κάποιος έλεγχο <laughs> και δεν επαληθευτεί αυτό το οποίο ζητάει στον έλεγχο, τότε θα πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να πληρώσει κάτι. <laughs> να κεράσει τον πρόεδρο. Άντε και τη γραμματεία. 61 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται δβ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DV5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές 68 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 71 υπέρ κατά αποχές ασάφεια έλεγχος 71 πιστεύω ότι απορρίπτεται πέρας 27-36 απορρίπτεται πράγματι 72 υπέρ κατά αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 76 και 77 ταυτίζονται ψηφί υπέρ κατά αποχές δεκτές δεβεφτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 εκπίπτει 81 ψηφι κατά αποχές. Έλεγχος στην 81. Η Abstimmung ist 33 33-29 γίνεται δεκτή. 82 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ είναι κομική αυτή η τροπολογία λέει ο πρόεδρος κατά αποχές δεκτή 85 υπέρ κατά αποχές δεκτή 86 υπέρ κατά αποχές δεκτή 87 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΔΕΒΕΝΕΑ υπέρ κατά αποχές δεκτή ...89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 2 υπάρχει αντίρρηση. Είπαμε μόνο για τη μία. Όχι κύριε Πρόεδρε, η ομάδα μου έχει αντίρρηση όπως είπα προηγουμένως και στην τρόπο, προφορική τροπολογία 2. Όχι για την 3, για την 1 και τη 2 μονάχα. 91 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 94 υπέρ κατά αποχές δεκτή 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβαστική 6 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 100 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 101 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 106, 107, 108, που είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές δεκτές προφορική 3 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή. <clears throat> Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ για την 130 <clears throat> θέλετε έλεγχο εντάξει έλεγχος για την 130 η 131 δεν έχει ψηφιστεί ακόμα λέει η γραμματεία στον πρόεδρο 130 είναι αυτή που θα ελέγξουμε 130 λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Έλεγχος για την 130. Der Antrag ist geschlossen. Äh, Ψηφοφορία έκλεισε 32-26 γίνεται δεκτή. 131 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές Ούτε και αυτό είναι σαφέ. Παρακαλώ, με, το, με ανάταση χειρών. Ψήφι υπέρ τη 131. Κατά. Αποχές γίνεται δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αν είσαι υπέρ ή κατά δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ κατά <clears throat> αποχές δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. <clears throat> 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 1. Μόνο για το ισπανικό ε, γλωσσικό κείμενο. 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 4 και 7 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 6 υπέρ κατά δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή το συνολικό κείμενο ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 59 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, τέσσερις αποχές. Herzlichen Glückwunsch. Συγχαρητήρια κύριε συνάδελφε. Κύριε Ταβάρες, έχετε το λόγο. Συγγνώμη, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι πάρα πολύ σύντομο. Είχαμε αυτό το περιστατικό με τι προφορικέ τροπολογίε, δεν θα τι διαβάσω αλλά θα διαβάσω ένα τμήμα τη ε, Προφορική τροπολογία υπαριθμών 2. Τονίζει την ανάγκη ε, συμφωνιών επανεστοχής για να αναφέρονται απαραίτητα υποχρεώσει σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε σχέση και με τα δύο μέρη. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους ότι ίσως μας εξέπληξε αυτή η αντίρρηση του ΕΛΚ να παρουσιαστούν οι προφορικές τροπολογίες και παραβιάστηκε η συμφωνία που είχαμε πριν, αλλά ήθελα να είμαι επίσημος και να καταγραφεί ακριβώς ε, σε τι έφεραν αντίρρηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω είπα και σε άλλε περιπτώσει, νομίζω ότι δεν είναι ιδιαίτερα σκόπιμο σε αυτή την Επιτροπή να φέρνει κανεί αντίρρηση στην παρουσίαση προφορικών τροπολογιών, αλλά θα ήθελα να πω στου συναδελφού ότι η ομάδα μου είναι πρόθυμη να συμβιβαστεί σε μια γενική συμφωνία που μπορούμε να συζητήσουμε στο διευρυμένο Προεδρείο και ε, να μην υπάρχει αντίρρηση από καμία ομάδα στις ε, προφορικές τροπολογίες. Απλώς εγώ ήθελα να σας πω ότι αν οι ομάδες σέβονται αυτή τη συμφωνία, τότε θα, και είμαστε, θα είμαστε και οι πρώτοι που θα τη σεβαστούμε. Σας ευχαριστώ. Κύριε Ταβάρες, όταν έχετε μια, ένα θετικό αποτέλεσμα και δεν υπάρχει καμία ψήφος κατά, θα πρέπει να είστε ευγνώμων στην Επιτροπή και να ξεχάσετε τα θέματα αυτά που σας οδήγησαν σε όργη. Ε, είναι, σχεδόν, είναι πολύ σπάνιο να έχετε μια έκθεση που περνάει χωρίς καμία ψήφο κατά. Περνάμε στην, στην έκθεση Ντόνσκης, ε, ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα μακρινάρι και χρειάζεται κάποια υπομονή από όλους μας. Πάμε. 60 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. 61 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. δεκτή. 62 υπέρ. Κατά αποχές Δεβένα, ΔΕΒ1 υπέρ. Κατά αποχές Δεβε ΔΕΒ2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 63 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 64 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σαφές. 67 υπέρ λέει ο πρόεδρος κατά αποχές απορρίπτεται. 68 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικά ελέγχουμε για την 69. Πέρας, σχεδόν πέρας, πέρας, 41 ψήφοι έναντι 17. Γίνεται δεκτή. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Φεμ 5 των γυναικών. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 73 υπέρ. Κατά Ούτε αυτό είναι σαφές. Απολύτως, αλλά σας ζητώ να συμμετέχετε στις ψηφοφορίες. 73. Λοιπόν, παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας και να μην καθυστερούμε. 73. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Και σας παρακαλώ και πάλι να συμμετέχετε στις ψηφοφορίες για να πηγαίνουμε πιο γρήγορα. Πέρας. 22 με 29 απορρίπτεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεκτή. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 80 σε δύο τμήματα. 79 πρώτα. Έλεγχος ηλεκτρονικός. Είναι τρίτη φορά. Πέρας ψηφοφορίας. Εντάξει, απερίφθη. 80. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 83. Υπέρ. Κατά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 97 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 96 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 98 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 100 και 101 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 110 και 111 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 112 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114, 115, 116 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 124. Υπέρ. 124. Κατά αποχές δεκτή. 126. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 128. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 129. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, 136. 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 137. Πέρας. με πολύ μικρή πλειοψηφία γίνεται δεκτή, 47-9. 138, 138 διορθώνει ο πρόεδρος, 138 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 139 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 140 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 141 και 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή 153 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 154 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται DV9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φεμ 11 υπέρ κατά και πάλι υπέρ φεμ 11 κατά αποχές γίνεται δεκτή 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 164 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος. Πέρα στις προφορίες 164 21-31 απορρίπτεται πράγματι. Κατά 65 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Εγκρίνεται. Κάποιοι κρατάνε το, κάποιοι κρατάνε το, τις ενδείξεις τους πολλή ώρα και εμπερδεύεται ο κόσμος. Λοιπόν, ήμασταν στην... Πού ήμασταν? 164. Όχι, ήμασταν στην Κόμες. 165 του λέει η γραμματεία του Πρόεδρου. Την ψηφίσαμε. Ωραία. 166. 6 μαύρο υπέρ. 166 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές. Δεκτή. 175. Άρχεται η ψηφοφορία, λέει ο πρόεδρος. Συμβιβαστική 7. Επαναλαμβάνει. Πέρας. 31-24 γίνεται δεκτή. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 178 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή 100 έλεγχος ψηφίσατε υπέρ πρέπει να πηγαίνουμε λιγάκι πιο αργά λέει ο πρόεδρος πέρας Απορρίπτεται πράγματι. 26 με 30. 181 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 182 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 184 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 187 υπέρ κατά δεκτή 188 υπέρ κατά αποχές 188 υπέρ και πάλι κατά αποχές δεκτή 189 υπέρ κατά αποχές δεκτή 190 υπέρ κατά αποχές δεκτή 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φεμ 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Φεμ 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεβε 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΤΒ4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ΤΒ5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 194 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 196 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 λέει ο πρόεδρος αλλά έχει εκπέσει. 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 203 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 6 έχει εκπέσει 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 208 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 211 υπέρ όχι δεν έχει γίνει δεκτή 209 ψηφίζουμε 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φεμ 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ναι, ήταν οριακό. Οι φιλελεύθεροι τι είπαν, ναι ή όχι. Έλεγχος για τη 215 τότε. «215. Έλεγχος ηλεκτρονικός». Πέρας. 30-26 γίνεται δεκτή 215. 2-14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.16 υπέρ. Κατά. Τι γίνεται, Άννα, ναι ή όχι λες τώρα. Υπέρ. Υπέρ. Υπέρ. Μα νόμιζα ότι λένε πάντα όχι. κρατά το χέρι τόση πολλή ώρα που να δίνει σήμα και στο ναι και στο όχι, και στο υπέρ και στο κατά και μπερδεύει την ψηφοφορία. Λέει στην αναγκόμη ο πρόεδρο. Δεκτή 216, Δεβε 7 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 9, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 221, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 2.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ κατά αποχές απο... εγκρίνεται Συμβαστική 10 είπε Κατά. Κύριε Ισηγητά. Θα ήθελα να φέρω αντίρρηση στην ε, προφορική τροπολογία. Έχω αντίρρηση λοιπόν. Ich stimme über Kompromiss 10 ohne den mündlichen Änderungsantrag ab. Wer ist dafür? Τροπολογία συμβαστική 10 χωρίς την προφορική τροποποίηση. Ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή χωρίς την προφορική τροποποίηση. Ερχόμαστε στη 235 υπέρ κατά αποχές δεκτή. ΦΕΜ 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒ 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 236 γέγλε υπέρ κατά αποχές πάλι 2.36 και πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.43 υπέρ κατά αποχές υπέρ είναι οι υπέρ εντάξει ωραία εγκρίνεται 2.44 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 2.46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.48 και 2.54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 12. Παρακαλώ, κύριε Ισηγητά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω να παρουσιάσω μια προφορική τροπολογία. από, ε, θέλουμε να λέμε the u based company και όχι Swedish finished company. Will er er äh, Ersetzen mit EU-based. Ja, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Er möchte konkreter werden. Hm. Συγκεκριμενοποιείται η τροπολογία έτσι. Ποιο είναι υπέρ τη συμβαστική 12 με αυτή την ε, τροποποίηση, την προφορική κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται λοιπόν με αυτή τη μορφή. Πάμε στη συμβαστική 13. Ψήφι υπέρ κατά αποχές 13 και πάλι ψηφίζουμε συμβαστή 13 ηλεκτρονικά πέρας Κάτι δεν πάει καλά σήμερα. Πού είμαστε? Είμαστε στη 250... 256 υπέρ. Όχι, όχι, λέει η γραμματεία. Α, ψηφίσαμε μόλις 13. 253 πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 258 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 260 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 261 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2.65 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.66 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 2.68 υπέρ. Σαν πρόσθεση στην 2.65 κατά αποχές απορρίπτεται. 2.69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 2.70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.75 και 2.85 μάλλον κατά αποχές απορρίπτεται. 2.80 υπέρ. Α, ήταν μαζί οι δύο αυτές, 2.75 και 2.80. 2.76 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 2.78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2,81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2,83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2,87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.90 υπέρ κατά αποχές <clears throat> δεκτή 2.91 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 2.92 υπέρ. Κατά αποχές. Δεν είναι σαφές. Απορρίπτεται. Λέω 2.93 υπέρ. Κατά αποχές. Παρακαλώ. Ήσασταν υπέρ. <clears throat> Εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 2.96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.97 2.97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.99 υπέρ κατά αποχές δεκτή 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.01 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.02 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.03 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.04 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.09 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.05 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.06 υπέρ Υπάρχει μια προφορική τροπολογία από τον κύριο Τέκεσ. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Σχετικά με τους πρόσφυγες λόγω κλιματικών συνθήκων, προτείνουμε αντί της προώθησης της δικαστικής νομιμοποίησης αυτών των κλιματικών προσφύγων να αντικαταστήσουμε τη φράση ως εξής. Καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μελετήσουν την έννοια του κλιματικού πρόσφυγα. Υπάρχει αντίρρηση, επομένως δεν μπορεί να ψηφιστεί. 306 χωρίς προφορική τροποποίηση. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 307 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 308 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 310 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 311 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται φεμ 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 312 υπέρ κατά αποχές δεκτή έλεγχος Μα οι σοσιαλιστές υπερψήφισαν. Όχι, λέει η κυρία Γκόμης. Όχι, όχι, όχι. Μα... 12 λέει ο πρόεδρος. Ηλεκτρονικά. <laughs> Απορρίπτεται. 24 με 26. 3-13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 3.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3.18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.19 υπέρ κατά αποχές δεκτή Δεκτή. Συμβαστή 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.20 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 3.27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 3.25 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Εκπίπτει ΦΕΜ 12, 326 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 328 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτό. 329 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 330 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 331 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3.34 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 3.35 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Όλες οι, οι τροπολογίες της Επιτροπής Γυναικών, η ΦΕΜ, από κοινού. Συμφωνεί. 2, 4, 6, 8, 10. Ψήφι υπέρ. Υπέρ. Χωρίς την 4 και χωρίς την 7. Φεμ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μα οι σοσιαλιστές υπερψήφισαν. Έλεγχος, έλεγχος. δύο έλεγχος. Μα αφού έδειξαν ναι, λέει ο πρόεδρος. Και όχι, όχι. Λοιπόν, πέρας. Απορρίπτεται. Φεμ 4 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Φεμ 7 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Φεμ 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 8 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Φεμ 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 3.36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.38 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.38 λέω πρώτος και πάλι κατά αν την ψηφίσαμε αυτήν 3.37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Μία τροπολογία του κυρίου Πέτερλε δεν μπορεί καταρχήν να απορρίπτεται, το ξέρω, 339. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 340 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 341 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3.43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.45 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3.46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3.48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Προφορική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 Συγγνώμη. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 354 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 358 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Ερχόμαστε στην 360. Όχι, εκπίπτει. 363. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 364 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 365 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 366 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ το πρώτο. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό. 360 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε τώρα στην ε, συμβαστική 19 έτσι δεν είναι ...370 εν μέρη. Ψήφι υπέρ. 370 δεν καλύπτεται πλήρω υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 375 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 376 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 379 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 380 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 382 υπέρ όχι εγκρίνεται εγκρίνεται 380 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 381 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 383 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 385 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 387 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 3, 88 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 389 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 490 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 391 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 392 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 393 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 394 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 395 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται εκπίπτει 397, 398 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 401 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 402 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 403 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή, 404 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Φεμ 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φεμ 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φεμ 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φεμ 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φεμ 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στην 2 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Φεμ 20 2. Φέμ 22 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ. Κατά. 4 υπέρ και πάλι. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Δεχτή. 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 7 και 8 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 9, 10 και 11 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτές. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 φεμ υπέρ κατά αποχές δεκτή φεμ 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται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 Wir haben es zu Ende mit 47 zu 0 47-0 γίνεται δεκτή η έκθεση. Συγχαρητήρια και Ντόλσκης. Wir kommen zum äh, Opinion Peterle. Και να περάσουμε τώρα. Στην... Έχουμε την τροποποίηση 1, εγκρίνεται, τροποποίηση 2, εγκρίνεται, τροπολογία 2, εγκρίνεται, του κ. Πέτερλου στο κείμενο του Πέτρελε 3 απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου του κυρίου Πέτερλε υπέρ κατά πέρας της ψηφορίας Μάλιστα. Έχουμε 50 ψήφους υπέρ, 2 κατά. Συγχαρητήρια. Και να περάσουμε τώρα στην έκθεση Σάρου Τσουβόλσκι. Λοιπόν, 2 εγκρίνεται. Τροπολογία 5 εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται και να περάσουμε στην 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ, όχι, 22, 22 λέει ο πρόεδρος, υπέρ κατά αποχές, 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στο τριστροπολογία 6 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29. Καταπίπτει, δεν είναι σωστό στον κατάλογο. 31 λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 33 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο του κειμένου αρχίζει η ψηφοφορία Πέρας. Σαράντα μία υπέρ, δύο κατά, έξι εποχές. Χαρητήρια. Σήμερα έχουμε ευρύτατες πλειοψηφίες της γενικές πληροφορίες, ψηφοφορίες και θα πρότεινα τώρα να περάσουν στο σημείο 9 της ημερησίας διάταξης γιατί ήρθε η κυρία Επίτροπος έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ανάπτυξη. Ποιο θα ασκήσει καθήκοντα Προέδρου. Θέλετε να προεδρεύσετε γιατί εγώ σε λίγα λεπτά πρέπει να φύγω. Oh, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Επιστρέψτε στις θέσεις σας. Έχω τη μεγάλη χαρά να υποδέχομαι την Επίτροπο την κυρία Γεώργιοβα, η οποία είναι αρμόδια για τα θέματα διεθνούς συνεργασίας, ανθρωπιστικής βοήθειας και αντιμετώπισης κρίσεων. και έρχεται να μας μιλήσει για την κρίση στην Συρία. Πρόκειται για μια σύραξη η οποία έχει μεγάλη σημασία για όλους μας και η οποία μας ανησυχεί βαθύτατα. όχι μονάχα το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στη Συρία, αλλά και τα ανθρωπιστικά προβλήματα που έχει προκαλέσει και τα θέματα ασφάλειας για τους ε, βρισκόμενους στη Συρία αλλά και σε αυτούς που βρισκόνται σε κατευλισμούς προσφύγων στην Τουρκία. Και επίσης υπάρχουν ενησυχίες σε σχέση με το περιβάλλον αυτής της κρίσης που μπορεί να επεκταθεί στο Λίβανο και ξέρουμε ότι και το Ιράκ σε κάποιο βαθμό έχει εμπλακεί σε αυτή την κρίση. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που η κυρία Επίτροπος είναι έτοιμη να κάνει μια δήλωση ενώπιόν μας. Πιστεύω ότι όλοι σας συμφωνείτε ότι έχουμε κάθε καθήκον να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση στη Συρία και κυρία Επίτροπε είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τις δικές σας εκτιμήσεις και τις ε, προτάσεις σας για το θέμα αυτό και κάνουμε τώρα μια κοινή συνεδρίαση με την ε, Επιτροπή ε, Ανάπτυξης. Θα ήθελα να ζητήσω από την κυρία Ζολή, την πρόεδρο της Επιτροπής Ανάπτυξης, να αναλάβει τα ηνία της Προεδρίας για την τρέχουσα συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, πρόκειται να μιλήσουμε για την πολύ σοβαρή κρίση που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή στη Συρία. Έχει πάνω από 30.000 νεκρούς και πάνω από 275.000 άτομα τα οποία εγκατέλειψαν τη Συρία. Και σήμερα αυτά τα άτομα βρίσκονται σε καταβλισμούς στο Λίβανο, στην Τουρκία, στην Ιορδανία και στο Ιράκ. Πραγματικά λοιπόν θέλουμε να ακούσουμε τι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πράξει για να ενισχύσει, να εξασφαλίσει μάλλον την ασφάλεια αυτών των προσφύγων που έχουν πάει σε χώρες που κινδυνεύουν να αποστοθεροποιηθούν, όπως η Ορδανία και ο Λίβανος. Κυρία Επίτροπε, σας δίνω αμέσως στο λόγο λοιπόν για να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ευγνωμών που έχω την ευκαιρία να ενημερώσω την κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών σε σχέση με την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, το τι πράττουμε και πώς βλέπουμε το μέλλον. 21 μήνες έχουν περάσει από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση χωρίς να έχει εξευρεθεί πολιτική λύση. Συνεχίζεται η εσωτερική μάχη, πλησιάζεται και ο χειμώνας και συνεπώς η ανθρωπιστική κρίση επιδεινώνεται και γίνεται τρομακτική πλέον θα έλεγα. Όπως είπατε κυρία Ζολή, πάνω από 30.000 άνθρωποι έχουν ήδη χάσει τη ζωή τους, πάνω από 2,5 εκατομμύρια και αυτό είναι υποτιμημένο στοιχείο, ε, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια 1,2 εκατομμύρια έχουν μετακυρηθεί εσωτερικά. Ακούμε πολλά για αυτούς που έχουν περάσει τα σύνορα, αλλά και οι εσωτερικές μετατοπίσεις σημαίνει ότι η δημόσια κτίρια που θα ήταν σχολεία τώρα έχουν ε, καταληφθεί από μετατοπιστέντες και έχουν μετατραπεί σε κατοικίες. Έχουμε 500.000 Παλαιστινίους πρόσφυγες στη Συρία και όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες τους εμπλέκουν στη σύραξη. Έχουμε και 100.000 πρόσφυγες από το Ιράκ στη Συρία και αυτοί βρίσκονται σε ιδιαίτερη, ιδιαίτερα δυσχερή κατάσταση γιατί δεν έχουν κοινωνικό ιστό στον οποίο να βασιστούν για βοήθεια. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσφύγων στις γειτονικές χώρες Τουρκία, Ιορδανία, Ιράκ έχει ξεπεράσει τους 222.000 και ενδεχομένως έχουμε και πολύ περισσότερους που δεν είναι εγγεγραμμένοι, που ζουν με την οικογένεια ή φίλους. Έχει κλιμακωθεί πολύ γρήγορα η βία από το καλοκαίρι. Από τότε που η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ταξινόμησε αυτή την σύραξη σαν εμφύλιο πόλεμο. Έτσι τη χαρακτήρισε. Αυτό το οποίο είναι πραγματικά τρομερό είναι ότι από τον Αύγουστο η κυβέρνηση έχει επιλέξει στρατιωτική, στρατιωτικές επιθέσεις βάλει τον αστικό πληθυσμό, τους πολίτες, ε, δεν εμπλέκονται τα στρατεύματα της Συρίας ε, σε ε, εμπλοκές από μακριά προκαλούν ε, από, από μακριά μάλλον επειδή έχουν μεγάλη υπεροπλία προχωρούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όταν πήγα σε ένα καταβλισμό προσφύγων στην Τουρκία ε, είχαν 20.000. Τον Ιούλιο φτάσαν στις 30.000. Τώρα έχουμε φτάσει σε 110.000 αυτοκαταβεβλισμό και δυστυχώς προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους ο αριθμός των προσφύγων σε αυτή την περιοχή θα ξεπεράσει τις 700.000. Και, αυτό, και μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια πολύ ευαίσθητη περιοχή και βεβαίως μπορεί να περάσει αυτός ο εμφύλιος πόλεμος και στους γείτονες. Τι κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μπλέξει στην τρομεκτική αυτή σύραξη. Ανθρωπιστική δράση, συντονισμός επιχειρήσεων και υποστηρίζουμε τα θύματα αυτής της σύγκρουσης. Χρηματοδότηση πρώτα απ' όλο Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη είναι ο μεγαλύτερος ανθρωπιστικός χορηγός. Έχουμε ήδη δώσει 250 εκατομμύρια ευρώ, 119 προέρχονται από την Επιτροπή και 96 από τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας μου, τον ανθρωπιστικό το Ανθρωπιστικό Ταμείο και τα υπόλοιπα από το Μηχανισμό Σταθερότητας και τους μηχανισμούς ε, καλής γυτνίασης σε συντονισμένο τρόπο. Αυτό είναι 47% ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας βάσει του, της καταγραφής από τον ΟΗΕ. Επίσης, έχουμε ενεργοποιήσει δύο φορές το μηχανισμό ε, προστασίας του πολίτη την πρώτη φορά για την Τουρκία και τη δεύτερη φορά το Σεπτέμβριο για την Ιορδανία. Όσον αφορά τώρα το συντονισμό, βεβαίως πρώτα απ' όλα συντονιζόμαστε στην έδρα μας με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με τους μηχανισμούς ευρωπαϊκής γετνίασης, με τα κράτη-μέλη που θέλουν να αναλάβουν κάποια δράση, αλλά ειδικότερα υπήρξαν πάρα πολλοί ενεργοί στη δημιουργία συνεκτικής ανταπόκρισης σε μια πολύ δύσκολη διεθνή κρίση μαζί με την ύπατη αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών και με και δημιουργήσαμε το φόρουμ, το ανθρωπιστικό φόρουμ στη Γενέβη με τη συμμετοχή όλων, της Ρωσίας, των Σύρων, των Ίδιων κτλ. για να συζητήσουμε αποκλειστικά για τα καταπήγοντα μέτρα, για την ανθρωπιστική κρίση, ώστε να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Έχει συνεδριάσει αυτό το φόρουμ πέντε φορές 9 Νοεμβρίου ξανά συνεδριάζει. Επίσης συντονιζόμαστε με τους συνεταίρους μας εβδομαδιαία. Οι συνθήκες μεταβάλλονται συνεχώς και πρέπει συλλογικά να είμαστε σε θέση να κάνουμε τη καλύτερη δουλειά που μπορούμε. Επίσης, παίξαμε έναν σημαντικό ρόλο σαν προωθητική δύναμη, ώστε να επισύρουμε την προσοχή στο γεγονός ότι η απουσία πολιτικής λύσης, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ο μόνος τρόπος τρόπος με τον οποίο ηθικά μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί σε αυτή τη σύραξη. Πρέπει να βοηθήσουμε την πρόσβαση για τις ανθρωπιστικές ε, ομάδες και να προωθήσουμε τον σεβασμό του, ε, του δικαίου του πολέμου ή ε, να μην δολοφονούνται παραδείγματος χάρη γιατροί και τα ασθενοφόρα να έχουν ελευθερία κινήσεων. Δεν μπορεί, είναι εύκολα τα πράγματα. Επισήραμε όμω διεθνή προσοχή στο γεγονό ότι ακόμη και σε ένα πόλεμο υπάρχει το δίκαιο του πολέμου το οποίο πρέπει να τηρείται. Έχουμε δημιουργήσει ένα σωστό έντονο παράδειγμα για την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία στην παροχή βοήθειας και θέλω να αναφερθώ στο πιο σημαντικό ζήτημα. Τι πετυχαίνουμε με τις προσπάθειες που έχουμε καταβάλει, με την χρηματοδότηση και με την υποστήριξη πολλών θέσεων. Σήμερα λοιπόν παρέχουμε βοήθεια σε τρόφες μας 1,5 εκατομμύρια ανθρώπους στη Συρία ε, επίγουσα ιατρική περίθαλψη επίσης. Έχουμε ξεκινήσει μία επιχείρηση για την παράδοση ε, σκηνών για το χειμώνα διαφόρων εξοπλισμών ε, στους πληθυσμούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα. Θερμάστρες κτλ. κλιμασκεπάσματα. Ε, έχω εδώ ένα χάρτη που πραγματικά σας δείχνει τι πραγματικά κάνουμε. η μισή μας βοήθεια πηγαίνει σε περιοχές που ελέγχονται από την κυβέρνηση. Το, η άλλη μισή πηγαίνει σε αυτές που αμφισβητούνται ή ελέγχονται από τους αντάρτες ή αλλάζουν χέρια συνεχώς. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι θέσεις που υποστηρίζουμε και ο συντονιστικός μας ρόλος ε, ε, δημιούργησε περισσότερες δυνατότητες για τις διεθνείς ΜΚΟ και για τον ΟΗΕ. Στους πρώτους μήνες της σύγκρουσης μόνο η πατιαρμοστία των προσφύγων και το Ερυθρό Σταυρός και η Μισέλνος μπορούσαν να παρέχουν βοήθεια. Σήμερα Όλες, ε, όλοι οι φορείς του ΟΗΕ εργάζονται μέσα στη Συρία και έχουμε 7 ΜΚΟ ε, που ε, και αυτές μπορούν να λειτουργήσουν μέσα στην Συρία, είναι ευρωπαϊκές. Έχουμε πάνω από 4.000 εθελοντές ε, πολύ διεθνές προσωπικό και κάποιο τοπικό προσωπικό που απασχολείται από τον ΟΗΕ και τις διεθνείς ΜΚΟ και αυτοί παρακολουθούν την εφαρμογή ε, των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Και πάνω σε αυτό το χάρτη που έχετε μπροστά σας βλέπετε με ποιους συνεργαζόμαστε και τι πράττουμε. Εκτός αυτών, η Συριακή, ε, πετύχαμε η Συριακή οργάνωση η Συριακή κυβέρνηση με συγχωρείτε να επιτρέψει σε τοπικές οργανώσεις να συμμετάσχουν σαν εταίροι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι δεν μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί παντού. Οι Σύριοι, ιδιαίτερα όμως οι νέοι, είναι πολύ, έχουν πολύ εθελοντικό πνεύμα και οι κοινοτικοί φορείς, οι επιτόποι, είναι αυτοί που ε, μπορούν περισσότερο να μας βοηθήσουν να πλησιάσουμε τον πληθυσμό. 60% των, ε, της χρηματοδότησης πηγαίνει στη Συρία, 40% στις γειτονικές χώρες, ιδιαίτερα στην, προς την Ιορδανία και το Λίβανο έχουμε έντονα το συνέστημα ότι αυτές οι χώρες πρέπει πραγματικά να βοηθηθούν για να φέρουν γιατί φέρουν ένα μεγάλο βάρος από αυτό το πρόβλημα. Δίνουμε και κάποια βοήθεια στην Τουρκία, μικρό κομμάτι. Δεν μπορέσαμε να επεκτείνουμε τη βοήθεια προς την Τουρκία λόγω του τρόπου με τον οποίο ε, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις της Τουρκίας είναι οργανωμένες. Είναι βασικά κυβερνητικές και δεν μας επιτρέπεται να δώσουμε χρήματα σε κυβερνήσεις. Ακόμη πρέπει να σας τονίσω ότι η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει σπουδαίο έργο βοηθώντας ε, τους ε, πρόσφυγες αλλά είναι και χώρα με περισσότερους πόρους από ότι ο Λίβανος και η Ορδανία γι' αυτό θεωρούμε ότι οι προτεραιότητες μας απευθύνονται περισσότερο σε αυτές τις δύο χώρες και όχι τόσο στην Τουρκία. Λοιπόν, όποιο και αν είναι το επόμενο σενάριο, ξέρουμε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες θα παραμείνουν πολύ υψηλές για μεγάλο διάστημα. Είτε συνεχιστεί, συνεχιστούν οι σειράξεις ή αν υπάρξει ένα ξεχύλισμα στην ε, περιοχή ε, είναι αρκετά ε, αρκετά τρομακτικό ενδεχόμενο ή ακόμη και αν υπάρξει πολιτική συμβιβαστική λύση, δηλαδή τα βρούνε οι διάφορες πλευρές πολιτικά και σταματήσουν να πολεμούν. Ήδη τα όσα έχουν συμβεί είναι τόσο σοβαρά που ό,τι και να συμβεί θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε βοήθεια. Προσπαθούμε βέβαια στο μυαλό μας να αξιολογήσουμε την κατάσταση, ποια είναι η χειρότερη κατάσταση για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Ε, και τα χρηματοδοτικά μας σχέδια για τον επόμενο χρόνο βασικά ευθυγραμμίζονται με όσα έχουμε πράξει φέτος. Δηλαδή αναμένουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση σε υψηλό επίπεδο. Έχουμε τρεις τώρα βασικές ανάγκες όσον αφορά τους επόμενους μήνες. Η πρώτη είναι ανησυχίες μάλλον, συγχωρείτε, τρεις βασικές ανησυχίες. Το θέμα είναι αν θα έχουμε πρόσβαση ε, προς αυτούς που έχουν ανάγκη λόγω της σύραξης, η οποία μετακινείται πολύ γρήγορα από το ένα σημείο στο άλλο. Καμιά φορά δηλαδή βρισκόμαστε παράλυτοι όσον αφορά την παράδοση της βοήθειας και γι' αυτό ε, πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και τις δύο πλευρές ώστε να σέβονται το δίκαιο του πολέμου. Επίσης ανησυχούμε πολύ για τα επίπεδα της χρηματοδότησης. Σήμερα η έκκληση του ΟΗΕ χρηματοδοτείται μόνο κατά το ίμιση και οι ανάγκες αυξάνονται. Υποστηρίζουμε λοιπόν προς όλους, ιδιαίτερα προς τους Άραβες αλλά και προς χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα, ότι χρειάζονται να κάνουν περισσότερο για τα ανθρωπιστικά άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα ανθρωπιστικά πιστεύουμε κατά τρίτο λόγο ότι ο μόνος τρόπος να λυθούν όλα αυτά είναι μια πολιτική λύση μετά από διαπραγμάτευση. Όσο δεν υπάρχει αυτή, μόνο στήριξη μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Όμως, χρειαζόμαστε μια πλατφόρμα συνένωση όλων των δυνάμεων για τη λύση του προβλήματος της Συρίας. Τώρα, πώς ακόμη μπορούμε να επεκτείνουμε την πρόσβαση, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα. Έχουν υποβληθεί τρεις προτάσεις μέχρι τώρα. Μία για ανθρωπιστικούς διαδρόμους, δύο για ζώνες προστασίας, τρίτη για ενισχυμένες διασυνοριακές παραδόσεις. Όσον αφορά τους ανθρωπιστικούς ε, διαδρόμους, κοιτάξτε που είναι οι σειράξει ε, στον, χάρτη. Από πού, πού λοιπόν θα φτιάξουμε αυτούς τους διαδρόμους, ποιος θα προστατεύσει αυτούς τους διαδρόμους, εφόσον δεν έχουμε ψήφισμα του ΟΗΕ, πώς ε, θα εξασφαλίσουμε αυτούς τους διαδρόμους και πώς θα ξέρουμε ότι ο διάδρομος αυτός χρησιμοποιείται μόνο ανθρωπιστικά και όχι για το λαθρομπόριο όπλων. Το ίδιο ισχύει και για τις ζώνες προστασίας. Ποιος θα τις προστατεύσει αυτές τις ουδέτερες ζώνες ας πούμε. Πώς ε, θα είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ό,τι έχουν δηλωθεί σαν και ακόμη, πώς θα ξέραμε ότι αυτές οι ζώνες δεν θα, θα οδηγήσουν στον διαμελισμό της χώρας, κάτι που είναι μεγάλος κίνδυνος για την Συρία, δυστυχώς. Διασυνοριακά τώρα. Προς το παρόν δεν υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις της διασυνοριακές, διότι μπορεί να είναι δύσκολη η πρόσβαση και περιορισμένη, αλλά την έχουμε μέσα στη Συρία. Και αν υποστηρίξουμε τις διασυνοριακές επιχειρήσεις, ε, θα, ε, θα κινδυνεύσουν οι ζωές των ε, εθελοντών στους ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Ήδη 13 έχουν πεθάνει και μπορεί να μην μπορέσουμε και να παραδώσουμε στους σωστούς πληθυσμούς, διότι για τη Συριακή κυβέρνηση είναι η διασυνοριακή μεταφορά παράνομη και μη επιτρεπόμενη. Συνεπώς δεν έχουμε ακόμη καμία ένδειξη ότι οι διασυνοριακές δραστηριότητες ε, είναι αποτελεσματικές. αυτή η βοήθεια κατά 50 με 75% δεν ξέρουμε που καταλήγει ε, όταν προέρχεται, ακολουθεί διασυνοριακή οδό. Του του λεχθέντος όμως είμαστε ανοιχτοί για οτιδήποτε θα μπορούσε να βοηθήσει τους πληθυσμούς, τον λαό, αρκεί να είναι λογικό και πρακτικό. Δεν υπάρχουν ε, πράγματα τα οποία μας σταματούν. Ο μόνος μας στόχος είναι τα θετικά αποτελέσματα. Τώρα, μετά από τρία χρόνια ως Επίτροπος πρέπει να σας πω ότι έχω δει πολύ δύσκολες επιχειρήσεις σε πολλά μέρη. Όμως αυτή είναι η πιο περίπλοκη όχι μόνο επειδή υποφέρουν περισσότεροι άνθρωποι, υπάρχουν και κρίσεις που αφορούσαν μεγαλύτερους πληθυσμούς, αλλά επειδή δεν υπάρχει προοπτική για να φτάσουμε στο τέλος της. Και ένα συμπέρασμα που σαφώς μπορώ να βγάλω είναι ότι κάθε φορά που εθελοτυφλεί ο κόσμος όσον αφορά την αποτυχία μιας χώρας ή τα προβλήματα μια χώρας, τα αποτελέσματα είναι πάντοτε δραματικά και σίγουρα η Συρία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Ευχαριστώ. Thank you so much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το δραματικό απολογισμό του τι συμβαίνει σε μια χώρα που βομβαρδίζει τον ίδιο του τον πληθυσμό. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο από τον ε, Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή έχουμε την Κερνίκα καθημερινά. Και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Πέτερινγκ. Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κυρία Γεώργεβα, έχω δύο ερωτήματα. Καταρχήν όμως θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τον ειλικρινή τρόπο και τη σοβαρότητα με την οποία έχετε αντιμετωπίσει το καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βοηθήσει τους πρόσφυγες στη Συρία, από τη Συρία στις γειτονικές χώρες. Έχω δύο ερωτήματα. Γνωρίζετε ότι δυστυχώς η Ρωσία και η Κίνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας έχουν εμποδίσει μια, ένα κοινό ψήφισμα. Εγώ θα ενδιαφερόμουν ιδιαίτερα να κατανοήσω ποια είναι η στάση της Ρωσίας και της Κίνας για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αν θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία Ξέρω ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό για τις κυβερνήσεις και των δύο χωρών αυτών. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα, εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε κάθε συμφέρον τις χώρες που διάκειται φιλικά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στην γειτονιά της Συρίας να τις υποστηρίξουμε και εδώ αναφέρομαι ιδιαίτερα στην Ιορδανία και στο Λίβανο θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για τις επιπτώσεις που προέρχονται από τα ρεύματα προσφύγων στην ε, ε Ιορδανία και στον ε, Λίβανο. Ήμουνα πρόσφατα στην Τουρκία και μίλησα και με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Ερντοάν, ο οποίος ήταν απόλυτα ανοιχτό για μια βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω βέβαια πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση στην Τουρκία αλλά θα πρέπει να δώσουμε, εφόσον το επιθυμεί, στην Τουρκία κάθε μορφή υποστήριξη. Μήπω θα μπορούσατε να μου δώσετε περισσότερε λεπτομέρειε για το θέμα αυτό. Και πάλι θα ήθελα να τονίσω την εκτίμησή μου για το έργο σα και το έργο των συνεργατών σα. Ευχαριστώ κύριε Ντεκάισερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε κυρία Γεωργίεβα. Συμφωνώ με το όσο είπε ο κύριος Πέτερινγκ για το εξαιρετικό έργο που γίνεται επί τόπου. Έχω δύο ερωτήσεις. Καταρχήν, η πρώτη φορά τις μορφές συνεργασίας που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των προσφύγων, των συμπροσφύγων με τις διάφορες κυβερνήσεις των χωρών υποδοχής. Στην Τουρκία, παραδείγματο χάρη, συμβαίνει το εξή. Ε, η Τουρκία ε, δέχεται να υπάρχουν ε, διεκταυλισμοί γιατί από ό,τι φαίνεται είναι πιο εύκολο να συγκεντρώνεται ο πληθυσμό στους καταβλισμούς. Ξέρω ότι η κατάσταση στο Λίβανο είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, πολύ πιο πολύπλοκη. Και αν η κυβέρνηση θέλει να διαχωρίσει αυτή την ε, πολιτική, την ιστορική της πολιτική από το τι συμβαίνει στη Συρία, πριν ε, λίγες ε, εβδομάδες δέχτηκε να βοηθήσει τους πρόσφυγες του Βορρά, αν έμεναν στα πλαίσια μιας οικογένειας, αλλά δεν ήθελε να ασχοληθεί με αυτούς τις ΜΕΚΑ. Έχει αλλάξει κάτι και αν η άρνηση ε, της ε, κυβέρνησης ε, του Λιβάνου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το Λίβανο. Θέλουμε να ξέρουμε αν υπάρχει μια υποχώρηση στο ζήτημα αυτό και αν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση κατορθώνει να έχει πρόσβαση σε όλους τους πρόσφυγες γιατί ε, διαφορετικά η πρόσβαση θα περιοριζόταν ε, σε Ισλαμικές ομάδες και θα ήθελα να ξέρω τι συμβαίνει στην Ιορδανία. Γιατί δεν έχουμε παντού την ίδια εικόνα και δεν μπορεί η δράση μας να είναι η ίδια παντού. Και κάτι ακόμη που θα ήθελα να σας πω. Είναι αλήθεια όταν ε, παρουσιάζεται ενώπιόν μας ε, η κυρία Άστον, ε, μπροστά στην αδυναμία που έχουμε και μπροστά στην τραγωδία που συμβαίνει, πραγματικά θυμώνουμε πάρα πολύ, είμαστε εξοργισμένοι, αλλά εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατορθώσετε, να διαφυλάξετε την ανθρωπιστική πτυχή ανεξάρτητα από το τι γίνεται σε πολιτικό επίπεδο, γιατί εδώ ε, πρέπει να υλοποιήσουμε ανθρωπιστικές δράσεις ανεξάρτητα από την πολιτική. Όταν μιλάμε για διασυνοριακές ε, επιχειρήσεις, ε, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί απέναντι στους πληθυσμούς και εγώ νομίζω ότι πρέπει να ασκηθεί πίεση και στους εταίρους σε χώρες όπως η Κίνα και η Ρωσία και πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλα μέσα πίεση πέρα από αυτά που χρησιμοποιούμε για να καταλήξουμε σε μια επίλυση αυτού του δράματος. Αλλά έχετε αρκετά κονδύλια και πού θα αναζητήσετε τα κονδύλια αυτά. Τρία άτομα έχουν ζητήσει ακόμη το λόγο και ξέρετε δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να περιοριστείτε στο 1,5 λεπτό. Η κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τα όσα μας είπατε και για το πολύ καλό έργο που υλοποιούν οι υπηρεσίες σας ε, στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτής της σύραξης. Θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω, υπάρχει και σύνορο με το Ιράκ. Κατανοώ ότι υπάρχει λιγότερη δραστηριότητα προς το παρόν στα σύνορα αυτά, αλλά υπήρχαν πρόσφυγες από το Ιράκ στη Συρία και από ό,τι κατάλαβα πολλοί πέρασαν τα σύνορα και πήγαν στο Ιράκ. Πώς λειτουργεί η σχέση μεταξύ των δύο χωρών και το Ιράκ με τη σειρά του διευκολύνει την ανθρωπιστική βοήθεια στη Συρία. Η άλλη ερώτηση που έχω θα ήθελα να συνεχίσω τόσο είπε ο κύριος Πέτερινγκ. Ε, είπατε ότι η Κίνα και η Ρωσία θα έπρεπε να συνεισφέρουν περισσότερο στην ανθρωπιστική προσπάθεια. Έχουμε κάποια αριθμητικά στοιχεία πόσο συνεισφέρουν σήμερα. Αλλά η πιο σημαντική συνεισφορά που θα μπορούσαν να δώσουν είναι πολιτική. Να μην ε, μπλοκάρουν τη δράση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, και έχουν ευθύνη γιατί είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και οι δύο. Είπατε ότι χρειάζεται πολιτική λύση. Εγώ σήμερα στην εφημερίδα διάβασα, τις Αμερικανικέ εφημερίδες διάβασα ότι οι Αμερικανοί διερευνούν νέες ε, δυνατότητες για ένα νέο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και μια νέα πλατφόρμα των ανταρτών ε, προωθείται και δίνεται περισσότερη σημασία στις δυνάμεις τις εσωτερικές παρά στις εξωτερικές. Στην προοπτική αυτή πώς πώς διαρθρώνετε τις ε, προσπάθειες των δικών σας υπηρεσιών με τη δράση, με την δραστηριότητα της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αρλάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε, και εγώ. Εκτιμώ τα όσα κάνετε και μας δώσατε μία ξεκάθαρη εικόνα της κατάστασης αλλά θέλω να ρωτήσω το εξή φαίνεται να κατανοείτε πολύ καλά ποιο είναι το κεντρικό ζήτημα εκεί. Πρόκειται για ε, μια στρατιωτική σύραξη, έναν φίλο πόλεμο και από τη μία πλευρά έχουμε όπλα να δίνονται στη μία πλευρά και ε, όπλα στην άλλη. Αναφερθήκατε στη βία που χρησιμοποιείτε και έχετε δίκιο. Έχουμε ένα ε, πολύ σκληρό καθεστώς που χρησιμοποιεί τα όπλα, αλλά πρέπει να ξέρετε και ότι ένα τμήμα των ανταρτών ε, είναι πολύ καλά οπλισμένοι και επίσης είναι κτηνόδης όπως και η κυβέρνηση σε πολλές περιπτώσεις. Και επίσης ε, ξέρετε ότι η Ρωσία και η Κίνο μονόπλευρα ε, παρέχουν όπλα και η κυρία Κλίντον είναι στην περιοχή προσπαθώντας να οργανώσει την ε, αντίσταση τους αντάρτες και είπε ότι αν αποτύχουμε αυτοί μπορούν να αποφασίσουν να δώσουν βαρύ οπλισμό στους αντάρτες. Γιατί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο απούσα πολιτικά, είμαστε εντελώς απόντες από όλα αυτά. Εμείς ε, κάνουμε πολύ καλή δουλειά, αλλά δρούμε ως ένα τεράστιο ερυθρό σταυρός. Λείπουμε όμως παντελώς από το πολιτικό σκηνικό. Γιατί δεν υποστηρίζουμε την εξέβρεση μιας πολιτικής λύσης εκεί, γιατί δεν υποστηρίζουμε παρκώς ε, το σχέδιο Ανάν και το σχέδιο Μπραχήμι, που φαίνεται να είναι τα μόνα συγκεκριμένα βήματα, οι μόνες συγκεκριμένες λύσεις ε, και για να επιληθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στην ε, ευρύτερη περιοχή, γιατί έχουμε και το θέμα της ανθρωπιστικής πρόσβασης. Κύριε Μπραντνερ, ναι, ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ, για τα όσα μας παρουσιάσατε και για όλο το έργο σας. Είναι καλά τα νέα. Είπε τώρα ότι υπάρχουν οργανώσεις σε τοπικό επίπεδο, γιατί ε, ο Ερυθρός Σταυρός ε, στη Συρία δεν θεωρείται ουδέτερος. Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τους Κούρδους. Ακούσαμε ότι για το κουρδικό τμήμα η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και υπάρχουν ε, πάρα πολλοί εσωτερικά εκτοπισμένοι σε αυτό το τμήμα της χώρας. Αλλά η υποστήριξη από τα έξω είναι πολύ αδύναμη και το χειμώνα θα έχουμε τραγωδία εκεί. Σε ποιο βαθμό είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Δεύτερο, είπατε ότι η χρηματοδότηση στον ΟΗΕ δεν έχει φτάσει ακόμη τα απαιτούμενα επίπεδα και αναφέρατε και άλλες χώρες. Αλλά ε, σε ποιο βαθμό συνεισφέρουν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο οι μεγάλε χώρε. Η Ουγγαρία, παραδείγματο χάρη. Θα μα ενδιαφέρει να μάθουμε κάτι τέτοιο. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Η κυρία Μουνή Δεουρκίσα. Ένα λεπτό έχετε. Μάλιστα, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Επίτροπε. Πολύ σύντομα θα ρωτήσω το εξή Πολύ πρόσφατα εκ μέρους ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών ε, από τους εξορισμένους Σύρους δημιουργήθηκε μια πρωτοβουλία για να φτάσει όλη η διεθνή βοήθεια στην Συριακή Αντιπολίτευση και στα επαλευθερωμένα εδάφη. Συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό κατά κάποιο τρόπο και ε, έχει έρθει σε επαφή με τη Χίλαρη Κλίντον ε, η οποία ε, ήταν και αυτή που σκέφτηκε αυτή την ιδέα. Μάλιστα σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Επίτροπος για να απαντήσει. Κύριε Γεωργίευ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, απαντήσω στις ερωτήσεις με τη σειρά που ακούστηκαν. Για τον κύριο Πέτερινγκ. Η συνεισφορά της Κίνας και της Ρωσίας σε σχέση με την οικονομική τους δύναμη και με, την ε, πολιτικά με το πολιτικό τους ε, στάτους είναι μικρή. Μέχρι τις 25 μάλλον, Σεπτεμβρίου, δεν έχω σημερινά δεδομένα, αλλά μέχρι τις τέλη Σεπτεμβρίου 2 εκατομμύρια δολάρια έδωσε η Κίνα και 9,5 εκατομμύρια η Ρωσία. Η Ρωσία επίσης ε, έστειλε ε, εκεί μια συνεισφορά σε είδος ε, αυτός ο μηχανισμός μοιάζει με τον δικό μα μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Αλλά νομίζω ότι πολλά περισσότερα θα μπορούσαν και θα έπρεπε να κάνουν. Πώς συμπεριφέρονται στα ανθρωπιστικά ζητήματα. Όταν ε, καλέσαμε το ανθρωπιστικό φόρουμ, το Συριακό Ανθρωπιστικό Φόρουμ, υπήρξε μία τάση να πολιτικοποιηθεί η συζήτηση και να αρχίσουν να δείχνουν για το ποιος φταίει. Αλλά πολύ γρήγορα κατορθώσαμε συλλογικά να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στις ανθρωπιστικές ανάγκες, στα δεινά του λαού. Και αυτό βοήθησε. Και πρέπει να πω ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε την επιρροή της για να πιέσει για περισσότερη πρόσβαση για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, ιδίως για τα Ηνωμένα Έθνη, για τις υπηρεσίες του ΙΕ. Αλλά δεδομένης ε, της ε, προοπτικής, πιστεύω ότι έχουν την υποχρέωση να δεσμευτούν περισσότερο για το θέμα της ατιμορρησίας και αν μου επιτρέπετε θα περάσω στα όσα είπε ο κ. Αρλάκη ε, υπάρχουν κτηνοδίες ε, σε όλες τις πλευρές. Ε, κάποιοι από τους αντάρτες προερχόνται από την Αλκάιτα, κάποιες, κάποια από αυτά τα από τρόπα εγκλήματα που έγιναν, έγιναν και από αυτού. Είναι θέμα μεγέθου. Η κυβέρνηση έχει καλύτερο εξοπλισμό και κάνει και πιο τρομακτικά πράγματα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει ότι τέτοια πράξεις δεν λαμβάνουν χώρα και από την άλλη πλευρά. όλοι οι διεθνείς πρωταγωνιστές θα έπρεπε να επικεντρωθούν στο σεβασμό του ανθρωπιστικού δικαίου. Αλλά υπάρχει πρόβλημα. Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο για τη Συρία και συνεχίσουμε να το λέμε αυτό όσο πιο δυνατά μπορούμε. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλουμε να υπαναχωρήσουμε <laughs> στις μέρες πριν τη δημιουργία υπο... του Ερυθρού Σταυρού και της υπογραφής των συμβάσεων της Γενέβης. προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση. Και λέμε, εντάξει, δεν μπορείτε να συμφωνήσετε επί τη πολιτική λύση, αλλά σα παρακαλώ να συμφωνήσετε για το σεβασμό των συμβάσεων των συνδικών τη Γενέβη. Και με τι δικέ σα παραμέτρου. Ξέρουμε ποιο μπορεί να συνομιλήσει με ποιον. Κάντε το. Αλλά δεν συμβαίνει ακόμη αυτό. Και σε σχέση με τις όμορες χώρες ε, και πόσο ε, τις θίγει όλη αυτή η κατάσταση στην Ιορδανία και το Λίβανο. Θα μπορούσε ο αντίκτυπος ε, να είναι καταστροφικός για την περιοχή. Και θα σας πω μια ιστορία που είναι όμως ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Όταν είχαμε τον βομβαρδισμό συγγνώμη, της βόμβας στο Λίβανο, τις ε, επόμενες ημέρες είδαμε το αντίστροφο κίνημα, δηλαδή μετακίνηση, να φεύγουν Σύριοι από το Λίβανο και να επιστρέφουν στη Συρία και να λένε ε, ότι στην πατρίδα μας είναι άσχημη κατάσταση, αλλά ίσως στο Λιβάνο να γίνει χειρότερη κατάσταση. 30.000 άτομα πέρασαν τα σύνορα από το Λιβάνο στη Συρία. Βέβαια, κάποιοι από αυτοί επέστρεψαν εκ νέου. Υποστηρίζουμε την Ιορδανία και το Λιβανό με ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και με άλλα μέσα που έχει η Κομισιόν στη διάθεσή της για την Ιορδανία. Αυξήσαμε την, ε, την οικονομική, γιατί ο αντίκτυπο στις χώρες αυτές δεν ε, ε, είναι μόνο ότι υπάρχει κίνδυνος διάχυσης, αλλά υπάρχει και σοβαρός αντίκτυπος στις οικονομίες τους. Γιατί ένας πόλεμος δίπλα σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου τουρισμός. Και για την Ιορδανία και σε ένα μικρότερο βαθμό και για το Λιβανό είναι σημαντική πηγή εισοδήματο. Και η Τουρκία δέχεται σοβαρέ συνέπειε. Οι γειτονικέ περιοχέ τη Τουρκία που είναι κοντά στη σύνορα και όπου υπάρχει πολύ θρησκευτικό τουρισμό γιατί έχουν ε, κάποια σημαντικέ κάποιες σημαντικές θρησκευτικές τοποθεσίες, ε, έχουν φυγεί τα μάλα. Ο τρόπο που σκεφτόμαστε την υποστήριξη είναι η εξή. Ε, θέτουμε προτεραιότητα στι πλέον ευάλωτε χώρε, την Ιορδανία και το Λίβανο και το Ιράκ. Και θα φτάσω στο πώ μπαίνει σε αυτή την εικόνα και το Ιράκ. Γιατί για την Τουρκία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, έχει ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα υποστήριξης, σε μια μεγαλύτερη κλίμακα. Γιατί η Τουρκία επιθυμεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φέτος δίνουμε 960 εκατομμύρια ευρώ υποστήριξη στην Τουρκία. Όχι λόγω της κρίσης, αλλά επειδή επιθυμούν να, ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα χρήματα αυτά, περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ ε, δίνονται στην Τουρκία για να χτίσει κέντρα υποδοχή προσφύγων για να διαχειρίζεται καλύτερα το πρόβλημα των προσφύγων. Έτσι λοιπόν, θα έλεγα ότι όταν ε, δούμε την ευρύτερη περιοχή, Δίνουμε προτεραιότητα στην Ιορδανία και στο Λιβάνο γιατί είναι πιο ευάλωτε οι χώρε αυτές. Αν ε, θέλετε μπορείτε να συγκρίνετε και το μέγεθο της οικονομίας ε, και το εισόδημα, το κατακεφαλή εισόδημα. Αλλά έχουμε δώσει και χρήματα στην Τουρκία και έχουμε ενεργοποιήσει το MIC. Βέβαια, μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και για τους πρόσφυγες στην Τουρκία μέσω του ΟΗΕ, της υπατσαρμοστίας για τους πρόσφυγες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο για το όσα είπατε ότι ε, δεν μπορούμε να έχουμε μέτρα που να είναι κατάλληλα για όλα, γιατί διαφέρουν οι συνθήκες σε διάφορες χώρες, στο Λίβανο. Η κυβέρνηση για διάφορους λόγους δεν ε, έχει ιδρύσει καταβλισμούς μέχρι τώρα. Ε, οι πρόσφυγες πηγαίνουν να ζήσουν με οικογένειες. Η Ορδανία έλαβε την απόφαση να οικοδομήσει ένα καταβλισμό, αλλά υπάρχουν και εκεί πολλοί που ζουν με οικογένειες. Η Τουρκία κυρίως βασίζεται βασίζεται στην ίδρυση καταβλισμών, αλλά έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Τουρκία, γιατί όταν ε, δημιούργησε τον πρώτο καταβλισμό για τους 10.000 ε, θα μπορούσαν να κάνουν περισσότερο και τώρα έχουν 110.000 και συνειδητοποίησαν ότι ο τρόπος που έχουν ε, οικοδομήσει τους καταβλισμούς μπορεί να είναι απαγορευτικός για τους ίδιους και ήδη υπάρχει αρνητική αντίδραση στον πληθυσμό. Ίσως ε, θα πρέπει να βασιστούν λοιπόν περισσότερο στην υπατήρβαστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες, ε, για τη διαχείριση των καταβλισμών, για να υπάρχουν καλές συνθήκες και για τους ανθρώπους που προσφεύγουν εκεί, αλλά και συστήματα οικονομικά. Εμείς ε, θέλουμε να παίξει ο ΙΕ ένα μεγαλύτερο ρόλο και γι' αυτό υπάρχει, έχουν και τις επαγγελματικές ικανότητες να το κάνουν και τους ενθαρρύνουμε να διερευνήσουν την κατάσταση τρόπον που δεν είναι σε καταβλισμούς, δηλαδή πρόσφυγες που ζουν με οικογένειες. Εμείς ε, δίνουμε χρήματα για προγράμματα που προσανατολίζονται προς την κοινότητα και θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμη περισσότερο αυτά τα προγράμματα. Έχουμε αρκετά κονδύλια. Δεδομένου του θέματος ε, της πρόσβασης, των πόσων μπορούμε να κάνουμε και της αποφασιστικότητάς μας να παρακολουθούμε τα όσα χρηματοδοτούμε, έχουμε τώρα χρήματα μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτή είναι η δική μας πρόβλεψη. Έχουμε αύξηση 15 εκατομμυρίων και θα φτάσουμε στο επόμενο οικονομικό έτος και θα χρηματοδοτήσουμε από τον προπολογισμό του επόμενου έτους. Συνεργαζόμαστε στενά με τον Επίτροπο φίλε και με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να διασφαλίσουμε ότι όλα όσα γίνονται είναι αλληλοσυνδεδεμένα. Έτσι λοιπόν είμαστε συλλογικά πιο αποτελεσματικοί. Αρκούν αυτά. Εγώ πραγματικά ανησυχώ ότι η Συρία όχι μόνο υποφέρει, υπάρχει και μια τεράστια σκιά σε άλλες κρίσεις. Δηλαδή υπάρχει ένα τεράστιος αντίκτυπος, γιατί όσο περισσότεροι άνθρωποι πλήττονται, τόσο μεγαλύτερες οι ανάγκες. Αλλά αναγνωρίζουμε πόσο μεγάλο κίνδυνο μπορεί να αποτελέσει η Συρία για την περιοχή και για την Ευρώπη και φυσικά δίνουμε προτεραιότητα στη Συρία και το ίδιο θα πράττουμε και του χρόνου. Και τώρα μάλλον είναι το κατάλληλη στιγμή να πούμε πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ζητήσαμε κονδύλια για τα επόμενα 7 έτη και ερχόμαστε εδώ να τη χρηματοδότηση. Γιατί αυξάνονται οι ανάγκες, αλλά οι πόροι μένουν οι ίδιοι. Και τελικά Η ανασφάλεια δεν μένει σε ένα σημείο, αλλά διαδίδεται. Και εμεί δεν είμαστε ικανοί να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Για το θέμα του Ιράκ. Αρχικά το Ιράκ δεν ήταν μεγάλη ανησυχία. Λόγω του πώς διαδίδεται η σύγκρουση, η σύρεξη, αλλά ήταν και επικοδομητική μάλιστα. Στις 26 Σεπτεμβρίου Κάλεσα μια άτυπη υπουργική συνεδρία στη Νέα Υόρκη. Όλοι ήρθαν. Όλες οι όμορε και το Ιράκ συμμετείχαν. Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλεία και η Ρωσία και η Κίνα, όλοι οι κύριοι δωρητέ και οι άραβε δωρητέ. <coughs> και εντυπωσιάστηκα γιατί στη συνεδρίαση αυτή ήταν πολύ επικοδομητική η θέση του Ιράκ. Αλλά ανησυχούν. Και φτάνω στο κουρδικό δεν είχαμε ανησυχήσει τόσο πολύ για το κουρδικό τμήμα, γιατί οι ανάγκε δεν είναι τόσο μεγάλε εκεί, αν το δούμε σχετικά το ζήτημα. Η Συριακή Κυβέρνηση, μιλάμε για 8,2 της επικράτειας. Έτσι λοιπόν η Συριακή κυβέρνηση τους έχει αφήσει να είναι κάπως μόνοι τους. Είναι δύσκολη πρόσβαση, ναι μεν, αλλά οι ανάγκες δεν είναι και τόσο μεγάλες όπως ε, σε άλλες περιοχές όπου έχουμε πιο αγριές μάχες. Και για το πώς θα προχωρήσουμε σε πολιτικό επίπεδο. Μία νέα απόπειρα να έχουμε ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη Συρία θα ήταν πολύ πρόσδεκτο. Στις συναντήσεις με τους Υπουργούς Εξωτερικών υπήρξε σχετικά ομόφωνη στάση για τη Συρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προχωρήσει περισσότερο από όλους για τις κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων και κυρώσεων ε, που θίγουν δικές μας χώρες, όπως η Ιταλία και η Ισπανία, λόγω της απαγορευσής να αγοράσουν πετρέλαιο από τη Συρία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια που μπορεί να επιφέρει αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου τη κυρία Άστον, αλλά τακτικά συνομιλεί με την κυρία Κλίντον. Πιστεύω ότι υπάρχει μια επικοινωνία σχετικά με το πώ μπορούμε να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα και έχουμε και δύο κράτη-μέλη που είναι μέλη του Συμβουλίου ασφαλεία. και αυτό δίνει ιδιαίτερο στάτου στην Ευρώπη. Τώρα, σε σχέση με το ποιο κάνει τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία στοιχεία του Σεπτεμβρίου. Περίπου 140.000 ευρώ. Μικρή συνεισφορά, αλλά σημαντική. Αν δούμε τα κράτη-μέλη μας, τα περισσότερα έχουν ήδη αναλάβει δεσμεύσεις. Αλλά πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Αυτό είναι σαφές. Νομίζω ότι αυτές ήταν οι κυρίε ρωτήσεις που ακούστηκαν. Περισσότερη πίεση για πολιτική λύση για, από όλους και από αυτό τον οίκο είναι ευπρόσδεκτη. Bene, ringrazio... Μάλιστα. Ευχαριστώ την Επίτροπο, την κυρία Γεωργίδα. ευχαριστώ και την ε, Πρόεδρο Ζολή. Σας ευχαριστώ για αυτή την ε, παθιασμένη παρουσίαση και σας εύχομαι καλή δουλειά, γιατί τη χρειαζόμαστε. Συνάδελφοι, έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Στρατηγική της Ευρωπαϊκή Ένωσης για το κεραίο της Αφρικής. Ε, ο εισαγητής είναι ο κύριος Τάνοκ, ο αγαπητός συνάδελφος. Αυτό το σημείο δεν μπορεί να μας απασχολήσει πάνω από 40 λεπτά. Να προχωρήσουμε ταχαίως. Και είναι η δεύτερη φορά που αντελάσσουμε απόψει για αυτό το θέμα, για τη στρατηγική για το κεράς της Αφρικής. Η έκθεση αποτελεί ευκαιρία για τη δική μας Επιτροπή να αξιολογήσει πώς ε, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχή, κυρίως ε, στις σχέσεις με τις σημαντικές χώρες της περιοχής αυτής και γύρω από την περιοχή. Το να έχουμε ένα κρέας της Αφρικής ε, σταθερό και ασφαλές είναι μια αναγκαιότητα που επιβεβαιώνεται και από τις πολυόριθμες τροπολογίες 215. Χωρίς χρονοτριβή, να δώσω το λόγο στον κύριο Τάνοκ. Σας παρακαλώ να μην μακρηγορήσετε. Το κέρας της Αφρικής είναι πολύ ενδιαφέρον μέρος. Το Σουδάν, η Σομαλία, η Ουγγάντα εξακολουθούν να είναι, έχουν σειράξεις, αντιμετωπίζουν προβλήματα στην Ερυθρέα, στο Τζιμπούτι έλλειψη ε, κράτος δικαίου, λαθρεμπόριο, έχουμε τους πολέμαρχους, την Αλκάιντα και στο ανθρωπιστικό επίπεδο πείνα. Πέρυσι τον Οκτώβριο η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέβαλε μία έκθεση στρατηγικής και πρόσφατα η Ένωση διόρισε δύο εκπροσώπους στο Σουδάν για να προχωρήσει ο διάλογος στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η σταθερότητα για την παγκόσμια οικονομία. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό και το κέρας της Αφρικής μπορεί πολλά να συμβάλλει για ολόκληρη την Ήπειρο. Το κέρας της Αφρικής είναι προβληματικό όσον αφορά τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Είχαμε εξερασία το 2009, λοιμό, πάνω από 3 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται επίγουσα βοήθεια στο κέρας της Αφρικής. Μαζί με αυτό έχουμε ασταθή δημοκρατία και κακές προοπτικές, ιδιαίτερα για τους νέους. Οι νέοι που μεγαλώνουν σε πόλεις σαν το Μογκαντήσου γνωρίζουν μόνο τον πόλεμο και τη βία. Δεν έχουν προοπτικές και όλα αυτά αποτελούν γόνιμο έδαφος για την εγκληματικότητα, την πειρατεία, το λαθρεμπόριο, την υποστήριξη της τρομοκρατίας και βεβαίως έχουν χάσει και πολλά οι εφοπλιστές και οι ναυτικοί που συνελήφθησαν σαν όμοιροι μαζί με τα πλοία τους. Ακόμη έχουμε, βλέπουμε ότι αυτές οι ομάδες των πειρατών έχουν εξελιχθεί πολύ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει και οικονομικά όποιο χρειάζεται. Όμως η πολιτική ηγεσία πρέπει να έρθει από τις χώρες της Αιθιοπίας, της Κένιας και της Ουγκάντας που δυστυχώς αποσύρθηκε την περασμένη εβδομάδα από αυτή τη διαδικασία. Ε, είχε προσφέρει στρατιωτική υποστήριξη για τη σταθερότητα στην περιοχή και είχε επίσης ε, βοηθήσει για το Μακαδίσου και το Κουτσμάγια. Έτσι μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι βασικά η σταθερότητα πρέπει να έρθει μέσω των Αφρικανών για τους Αφρικανούς. Έχουμε και εκπαίδευση προσωπικού στην Ουγγάντα. Αυτή η στρατηγική θα συνεχιστεί συνεχίζοντας με το πρόγραμμα Νέστορ για την ανάπτυξη μιας αστυνομίας και θα προχωρήσουμε και στο Τζιμπουτί. Ακόμη χρειαζόμαστε και συντονισμό μεταξύ διακυβερνητικών μηχανισμών που μπορούν να παίξουν ε, περιφερειακό ρόλο για την καλή διακυβέρνηση. Η την πόρη είναι πολύ σημαντική. Έχουμε διαπραγματεύσεις και έχουμε και φράγματα στον ήλο το οποίο προχωράει. Ακόμη είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα στρατεύματα των Αφρικανών μπορούν να συνεργαστούν για να πετύχουν ε, το κοινό στόχο ακόμη μπορούν να προωθήσουν δημοκρατικές, δημοκρατική οργάνωση και δικαστικούς φορείς. Το Σουδάν ειρηνικά χωρίστηκε στα δύο και η δημοκρατία, η σταθερότητα θα υλοποιηθεί κάποια μέρα για όλους. Σαν εισηγητής μου έχουν υποβληθεί πολλές τροπολογίες, 215 μάλιστα, και αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέρονται οι συνάδελφοι για αυτό το θέμα. Όμως δεν είναι η πρόθεσή μου να επικεντρωθώ στα θέματα τα περιβαλλοντικά ή ανθρώπινα δικαιώματα. Βεβαίως θα ασχοληθούμε και αυτά. Όμως δεν θέλω να ανατρέξω στο παρελθόν, ιδιαίτερα όσον αφορά τις σχέσεις με την Αιθιοπία. Πρέπει να αφήσουμε την κυβέρνηση εκεί να προχωρήσει πρώτα. Εδώ μιλάμε για στρατηγική, ασφάλεια και οικονομικά θέματα σε αυτή την έκθεση. Γι' αυτό μπορούμε να πετύχουμε κάποιους συμβιβασμούς με συναδέλφους και ε, ε, έχουμε μία συνάντηση στο Στρασβούργο στην επόμενη Ολομέλεια να συναντηθούμε οι συγητές μαζί με τους σκιώδεις ώστε να μπορέσουμε να συντάξουμε κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες ε, για να ενοποιήσουμε τις διάφορες απόψεις. Αλλά είμαι τώρα στη διάθεση των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Χίλια ευχαριστώ. Να περάσουμε αμέσω στους συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Καταρχήν, συνάδελφος Βέντσον. Δύο λεπτά έχετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για αυτή την πλήρη παρουσίαση. Εγώ δεν χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Προφανώς υπάρχει και ηθική υποχρέωση και το επανέλαβε ο κ. Στάνο και ηθική υποχρέωση για όλους εμάς. Έχουμε δεσμευτεί για να εξεύρουμε συμβιβασμούς, συμβιβαστικές τροπολογίες για τη διατύπωση προκειμένου να υπερασπιστούμε τις θεμελιώδες ελευθερίες και προκειμένου όλοι οι πολίτες να ε, δουν τα δικαιώματά τους και την αξιοπρέπειά τους να γίνονται σεβαστά. Έχουμε και τις ε, χριστιανικές ε, ομάδες που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δυστυχώς καταπατούνται τα δικαιώματά τους από τον Ελένα και αυξανόμενο Ισλαμισμό. Θα πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε για να γίνονται σεβαστές οι θεμελιώδεις αρχές. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το επαναλάβουμε αυτό. Εδώ στην ΑΦΕΤ και μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να εξεύρουμε μία λύση για να προωθήσουμε αυτή την προβληματική. Τώρα υπάρχει μία νέα αισιοδοξία απέναντι στην Αφρική και απέναντι στη συγκεκριμένη περιφέρεια της Αφρικής. Η Ευρώπη ίσως ε, να μπορεί να ελπίζει σε καλύτερα αποτελέσματα σε σύγκριση με τα όσα έγιναν τα περασμένα έτη. Και η Σομαλιλάνδη αναφέρεται ως ένα καλό παράδειγμα. Θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτή τη χώρα να γίνει ανεξάρτητη Ο τρόπος που καθορίστηκαν τα σύνορα στην Αφρική πραγματικά είναι αμφισβητήσιμος. Για να το πω ευγενικά, θα μπορούσαμε να σκεφτούμε μια Σουμαλιλάνδη που να είναι ελεύθερη και ανεξάρτητη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Μουνίσο, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι 215 τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στην τροπολογία αυτή μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μια ευρύτερη προοπτική και εικόνα για τη σημασία της περιοχής και τον ρόλο που παίζει. Η εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να είναι μονάχα τα θέματα της ε, ασφάλειας, ούτε πρέπει να είναι τμήμα σταυροφορίας και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ευρύτερο τοπίο. Οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει τα μέλη της ομάδας μου νομίζω ότι εμπλουτίζουν την έκθεση του κυρίου Τάνοκ. Αναφέρονται καταρχήν στα γεγονότα που ακολούθησαν μετά από την παρουσίαση του πρώτου σχεδίου εκθέσεως. Στην Αιθιοπία ο θάνατος του πρόεδρου Φενάουι έχουμε καταθέσει τροπολογίες σχετικά. Επίσης, στη σύγκρουση μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας κάνουμε μία μνήα στο ψήφισμα ΟΗΕ, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τον Ιούλιο και τις προσπάθειες του ειδικού εισηγητή σε σχέση με το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Υποστηρίζουμε τροπολογίες οι οποίες αναφέρονται στη νέα συμφωνία που έχουν υπογράψει δύο χώρες και που επιτρέπει την ε, συνεργασία για να αντιμετωπιστούν τα μεταναστευτικά ρεύματα από το νότο προς το βορρά. Επίσης, εμείς υποστηρίζουμε την ε, συνέχιση της Aerofor και, της, ε, και του... της επιχείρησης Αταλάντα βάσει και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Μάιο του 2012 για την πειρατεία. Επίσης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι η πρότασή μας για τον έλεγχο των ε, εταιριών ιδιωτικής ασφάλειας έχει γίνει δεκτή από τον εισηγητή στην τροπολογία 90. Θεωρούμε ότι η δική μας τροπολογία 112, η οποία ζητά ένα κώδικα δεοντολογίας για αυτές τις ευαγείς υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας, είναι καλύτερη από αυτή του εισηγητού και περιμένουμε να βρούμε και μια συμβασική λύση για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την Σομαλία, υποστηρίζουμε την επιχείρηση εκπαίδευσης δυνάμεων ασφαλείας στη Σομαλία, και κάποιες πολιτικές ομάδες όπως οι πράσινοι έχουν καταθέσει τροπολογίες κατά αυτή τη ε, επιχείρηση που θεωρούν ότι είναι παρέμβαση εσωτερικά της Σομαλίας. Εμεί όμω υποστηρίζουμε τη συνέχεια αυτή τη ε, επιχείρηση για τον έστωρα και την υποστήριξη των ναυτικών ικανοτήτων και της ε, των ακτοπλοϊκών δυνάμεων. Υποστηρίζουμε και εμείς την απόφαση παριθμών 90 και 100. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ μονάχα σε δύο ακόμα θέματα. Στα θέματα ασφάλειας έχουμε εισαγάγει μια σειρά από τροπολογίες για την κατάσταση επίση των εκτοπισμένων εσωτερικά και των προσφύγων, που είναι σημαντικό θέμα. Έχουμε τονίσει επίση την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία με το Διεθνέ Ποινικό Δικαστήριο και θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα τη παράνομη πώληση ελεφαντοστού και την χρηματοδότηση με αυτού του τρόπου των πολεμάρχων στην περιοχή αυτή. Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει μια διαδικασία ανάλογα με τη διαδικασία του Κίμπερλε για το ελεφαντόδοτο και έχουμε φυσικά και το ψήφισμα για τη Σομαλιλάνδη που θα συζητήσουμε εν καιρό. Ευχαριστώ. Μπουτικόφερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ σε τρία σημεία. Σε ό,τι αφορά την πειρατεία, η δική μας θέληση είναι ότι η κυρία Άστον θα ακούσει καλύτερα τις συμβουλές που μας έδωσε ο Τζακ Λάγκ, ο ειδικό σύμβουλος του ΟΗΕ για τα θέματα πειρατείας, που αναφέρθηκε σε μια προσέγγιση για την ποινική δικαιοσύνη, για την αντιμετώπιση της πειρατείας. Ελπίζω θα μπορέσουμε όλοι να πορευτούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μια δεύτερη παρατήρηση σε ό,τι αφορά τη Σομαλία και τις γειτονικές της χώρες. Εγώ δεν θεωρώ ότι μια σειρά από μονομερείς περεμβάσεις όπως υπήρξε στο παρελθόν είναι χρήσιμες. Πιστεύω ότι αντίθετα εμείς θα πρέπει να τονίσουμε ότι από τη μία πλευρά, όπως λέει ο κύριος Στάροκ, θέλουμε μια αφρικανική ο κυριος Στάνοκ, αλλά αυτή η λύση θα πρέπει να έχει συλλογικό χαρακτήρα. Τρίτον, έχουμε μονάχα τον κύριο Ρόντο, Ρόντος ως ειδικό εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή θα ήταν χρήσιμο όμως να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπάνω για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο συντονισμό τη λεγόμενη <clears throat> συνολική προσέγγιση για την οποία πάντα εμείς αναφερόμαστε. Δεν πρέπει ο κ. Ρόντος μονάχα να είναι ο αρμόδιος για τα θέματα της ΚΕΠΑ, αλλά θα πρέπει να αναλάβει και την ευθύνη για τα περαιτέρω μέτρα τα οποία αντιμετωπίζει, τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να λάβει μέρος στις διαπραγματεύσεις με τους γείτονες της Σομαλίας και τη διαμεσολάβηση μεταξύ αντιμαχωμένων πλευρών. Ελπίζω λοιπόν ότι αυτά θα μπορέσουν να ληφθούν υπόψη. Σας ευχαριστούμε και που ήταν συλλοπτικός. Κατόπιν κυρία Γκόμες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Τόνατ για το αρχικό σχέδιο. Είμαι από εκείνου που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε απλά να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο κέρα της Αφρικής απλώ με την προσέγγιση της ασφάλειας. Χρειαζόμαστε κράτος δικαίου, διακυβέρνηση, και θέλουμε να ασφάλεια βεβαίω και θέλουμε να καταπολεμήσουμε την πειρατεία για την τρομοκρατία. Και όλα αυτά σημαίνουν ότι χρειαζόμαστε μια σοβαρή προσέγγιση και όχι αυτή που είχε η Ένωση προς τους εταίρους της περιοχής. Εφόσον δεν υπάρχει παροχή ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατίας λοιπά στις χώρες τους, πώς μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά ενισχύουν τους τρομοκράτες, διότι υπάρχει αυτή η ιστορία της περιοχής που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Ακόμη πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε την Αιθιοπία. Είναι στο κέντρο του κέρατος. Και ο θάνατος του Πρωθυπουργού Ζνάουελ ανοίγει βεβαίως ευκαιρίες, αλλά πρέπει να δεσμευτούμε και να υποστηρίξουμε τις δυνάμεις και ο νέος πρωθυπουργός ο οποίος έχει κάποιες δυσκολίες να ενισχύσει την εξουσία του σε σχέση με την παλαιότερη γενιά να μπορέσει αυτός να προχωρήσει σε ένα άνοιγμα. Είναι, δίνουμε πολλή ενίσχυση, πολλή βοήθεια βάσει της συμφωνίας Σκοτ, Σκοτονού αλλά έχει χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές. Αυτή είναι δουλειά για τις ευρωπαϊκές ΜΚΟ βεβαίως, αλλά πώς μπορεί αυτός να παρέχει κράτος δικαίου και ασφάλεια και δεν συμμαζεύεται στη γειτονική περιοχή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι η έκθεση αυτή μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Συμφωνώ για το ρόλο που μπορεί να παίξει ο κύριος Ρόντος Πρόσωπο μας, αν υιοθετήσει μια ευρύτερη προσέγγιση. Και θα ήθελα ακόμη να προσθέσω ότι ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα είναι η σύγκρουση μεταξύ Αιθιοπίας και Ερυθρέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα βάζει όλα κάτω από το χαλί και δεν κάνει τίποτα αντί να φέρνει αποτελέσματα στην περιοχή ρυθμίζοντας αυτή τη σύγκρουση. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Τόμας Φωνχάντελ από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, παρακαλώ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Πού είστε? Εδώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ε, λέγομαι Τόμας Φωνχάντελ, είμαι από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Λυπάμαι που ο διευθυντής μου Κοντερβάκτορ ήταν εδώ προηγουμένως, αλλά δεν μπόρεσε να μείνει, σας ζητά συγγνώμη, θα είχε μιλήσει εκείνος. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία, θα είμαι πολύ σύντομος. Χαιρόμαστε που η ΑΦΕΤ ασχολείται με αυτό το θέμα, είναι πολύ επίκαιρο και η έκθεση και το σχέδιο ψηφίσματος, διότι το στρατηγικό πλαίσιο για το κέρας της Αφρικής που υιοθετήθηκε πέρυσι αναθεωρείται τώρα μετά ένα χρόνο μετά την έγκρισή του, δηλαδή φέτος τον Νοέμβριο και βεβαίως μπορεί σίγουρα να υποφεληθεί από τις απόψεις, τις ιδέες και τις συζητήσεις που έχετε. Δεν έχω πολλά να προσθέσω, θα ήθελα μόνο να πω ότι η Κάθριν Άστον πράγματι έχει υπογραμμίσει σε πρόσφατο σεμινάριο επικεφαλής ε, αντιπροσωπιών κρατών ε, έχει, έχει τονίσει πρόσφατα το στρατηγικό στόχο και την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση που προτείνουμε στις ανασκοπήσεις που κάνουμε προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όλους τους μηχανισμούς που είναι στη διάθεσή μας και όλους τους συμβάλλοντες Έχουμε κατά νου βεβαίω τι αποστολέ που πραγματοποιούμε και τα κράτη-μέλη. Ένα σχόλιο θα ήθελα ακόμη να κάνω. Η Κένια παίζει σημαντικό ρόλο και έχει εκλογές το 2013 αυτές σίγουρα θα επηρεάσουν ολόκληρη την περιοχή. Βεβαίως η υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας να παρακολουθήσει τα θέματα, να βοηθήσει στην οριστικοποίηση της έκθεσης. Είμαστε γενικά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Τα συμπεράσματα στον συγγήτη. Παρακαλώ κύριε Τάνοκ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους συνοδέλφους που είχαν καλά λόγια για την έκθεσή μου και τις υποστήριξαν. Είναι, δύσκολος, είναι δύσκολο το θέμα για μια σύντομη έκθεση. Όπως σας είπα, επικεντρώνομαι βασικά στην περιοχή όσον αφορά την ασφάλεια, τα οικονομικά κτλ. Βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλέ άλλε πτυχέ και θα μπορούσε κανεί να συντάξει ολόκληρο βιβλίο, όχι απλώ κοινοβουλευτική έκθεση. Βεβαίω ε, το πιο λεπτό θέμα είναι στην Ερυθρέα. Υπάρχουν ε, διαβολικά θέματα που εξελίσσονται εκεί. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ βεβαίω σαν Βρετανός υποστηρίζω τη Σομαλιλάνδη και την αναγνώρισή της σαν ανεξάρτητη χώρα. Προσωπικά λοιπόν και η ομάδα μου θα υποστηρίξουν την τροπολογία σας προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά στο σχέδιό μου αναφέρω ότι ποια είναι τα θέματα που ενδιαφέρουν ειδικότερα την κυβέρνηση της Σομαλιλάνδης. Κύριε Λουκίζα, ήσασταν τόσο τηλεγραφική, ήδη δεν μπορούσα να τα σημειώσω όλο, όλα. Ναι, μιλήσατε για το ελαφαντοστούν. Ευχαρίστω να μιλήσω για τις, τα είδη που κινδυνεύουν. Χαίρομαι που οι σοσιαλιστές συμφωνούν για την επέκταση της εντολής του ΡΙΜΑΝΤ όσον αφορά τώρα την ιδιωτική ασφάλεια έχουμε πολλές ασφαλιστικές εταιρείε στο Λονδίνο και στη Βρετανία γενικά θα κοιτάξω τις τροπολογίες 100 και 112 με ενδιαφέρον θα προσπαθήσω να βρω ένα συμβιβασμό δεν είμαι υπέρ των υποχρεωτικών ε, διατάξεων. Είμαι υπέρ του κώδικα δεοντολογίας σε κάθε κλάδο. Ε, ακόμη δεν έχει υπάρξει πειρατεία σκάφους, ε, πλοίου μάλλον, όταν συνοδεύεται από ενόπλους. Κύριε Μπουτσικόφ, όσον αφορά την εντολή προς τον κύριο Ρόντο. Βεβαίως αυτό ξεπερνά το έβρος αυτής της έκθεσης, διορίζεται από το Συμβούλιο. Νομίζω ότι ε, του έχει δοθεί μια ευρία εντολή για την περιοχή. Τον έχω συναντήσει τον κύριο. Ε, προσπαθεί να φέρει αντιμαχόμενα μέρη μαζί, αλλά η εξουσία του, εν πάση περιπτώσει, προέρχεται από το Συμβούλιο. Ε, στους τομείς που μας ενδιαφέρουν και όσον αφορά την διαμεσολάβηση μεταξύ περιοχών, κυβερνήσεων κτλ. Σομαλία, Ερυθριά, Σομαλιλάνδη κλπ. Ξέρω ότι είχε ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα της Ερυθρέας ε, και ε, ήταν πολύ προσεκτικό στην διατύπωση που ήθελε να έχω. Κυρία Γκόμες, Σύμφωνα με πολλά από αυτά τα οποία είπατε, αλλά αυτή η έκθεση βασικά ενδιαφέρεται για την CFSP. Βεβαίως θα υπάρξουν και άλλα στοιχεία τα οποία θα ενταχθούν για να μπορέσει να γίνει η ειρηνική περιοχή ε, το κέρας της Αφρικής κάτω από καλή διακυβέρνηση. Όσον αφορά το σχολείο σας για την Ίγκα, το σημειώνω, αλλά δεν μπορούμε, θα χρειαστεί να συνεργαστούμε, δεν μπορούμε να αναδομήσουμε την αρχιτεκτονική της περιοχής. Πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτά που έχουμε. Η Αιθιοπία βεβαίως είναι ε, κεντρικό θέμα για την περιοχή, είναι στρατηγική σχέση, αλλά προτιμώ να αντιμετωπίσουμε τη νέα κυβέρνηση με ευγένεια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι τελειώσαμε και θα έχουμε και συνεδρίαση με τους Σκιώδης στο Στρασβούργο στην επόμενη ολομέλεια. Ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Το επόμενο σημείο αφορά μια ενημέρωση από τον κύριο Παύλ Κόβελ σχετικά με την αποστολή εκλογικών παρατηρητών στις βουλευτικές εκλογές της Ουκρανίας στις 28 ε, Οκτωβρίου του 2012. Στις 20 Οκτωβρίου έλαβαν χώρα κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ουκρανία θεωρήθηκαν πραγματικό τεστ για τη δημοκρατία στην Ουκρανία και συζητήθηκαν εκτενώς πριν από την εκλογική αναμέτρηση. Έγινε μάλιστα στις 11 Οκτωβρίου και ένα workshop από μας. Αυτές οι εκλογές θεωρήθηκαν τόσο σημαντικές ε, που έστειλε η Ευρωπαϊκή Ένωση 15 παρατηρητές ε, στην αποστολή, μια μεγάλη αποστολή και ε, έστειλε στις αρχές Οκτωβρίου και μια προεκλογική αποστολή στο Κίεβο. Επικεφαλής ήταν ο κύριος Πάβελ Κόβελ, ο οποίος συμμετέχει και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνεργασίας με την Ουκρανία. Συνήθως η αποστολή αυτή ήταν τμήμα της Διεθνούς Αποστολής Εκλογικής, Εκλογικών Παρατηρητών. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από την έλλειψη ισότιμων κανόνων κυρίως λόγω της κατάχρησης των διοικητικών πόρων, την έλλειψη διαφάνειας, την αναμέτρηση ε, της εκλογικής εκστρατείας και μειωμένη έλλειψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Επίση, τα συμπεράσματα λένε ότι οι ψηφοφόροι ε, γενικά μπορούσαν να επιλέξουν ε, μεταξύ των κομμάτων ε, υπήρξε ηρεμία τη μέρα της εκλογής και τα γενικά αποτελέσματα θεωρούνται θετικά. Υπήρξε έλλειψη όμως της αφήνειας, τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη.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 Προέδροβα είχα μαζί μου τον κύριο Γκάλερ, τον κύριο Χουάν Φερνάντε Λόπες Αγγιλάρ και την κυρία Ρεμπέκα Χάρμς. Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας μας πήγε στο Κίεβο. Δεν μπόρεσαμε όλοι μας να μεταβούμε εκεί. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ότι η παρουσία μας στην προεκλογική περίοδο ήταν πολύ σημαντική, γιατί είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με εκπροσώπους πολλών πολιτικών κομμάτων, αλλά και πολλών φορέων της κοινωνίας των πολιτών. Συζητήσαμε και με τον κύριο Βίνσκι και με τον επικεφαλής της ε, αποστολής του Ιδρύματος για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η συνεργασία μας ήταν λοιπόν πολύ θετική με όλους αυτούς τους φορείς. Κάνουμε λοιπόν αυτή την αναγνωριστική ε, αποστολή η οποία προηγήθηκε της ίδιας της παρακολούθησης των εκλογών. Δώσαμε μία αναφορά για τα θέματα αυτά στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και συμμετέσχαμε επίσης και σε ένα σεμινάριο σε σχέση με την παρακολούθηση των εκλογών. Θέλω να σας υπενθυμίσω ποια είναι τα βασικά μας συμπεράσματα. Όταν έλαβα το λόγο προηγουμένως στην Επιτροπή μας, τόνισα ότι ο νέος εκλογικός νόμος ο οποίος έγινε δεκτός και από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση το 2011, εισήγαγε ένα μεικτό σύστημα ψηφοφορίας. Σήμαινε αυτό στην πράξη μισές έδρες στο Ανώτατο Συμβούλιο κατανέμονται βάσει ενός πλειοψηφικού συστήματος και θεωρούσαμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε προβλήματα. Δυστυχώς επαληθεύτηκε η πρόβλεψή μας. Πρέπει να σας υπογραμμίσω ότι δεν λειτουργήσαν σωστά οι εκλογικοί κατάλογοι στην ε, Ουκρανία και δεν εφαρμόστηκε και η ίδια η νομοθεσία με κάποια σαφήνεια, κάτι το οποίο είχαμε αναφέρει σε σχέση και στο παρελθόν σε σχέση με τις εκλογικές επιτροπές. Υπήρξαν πλασματικά κόμματα. Και βάσει του νέου εκλογικού νόμου στην Ουκρανία αυτά τα πλασματικού χαρακτήρα, τα κόμματα αυτά είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συμμετοχή στις εκλογικές επιτροπές, ενώ πραγματικά κόμματα όπως το Σφόμποντα και το Ούνταλ που είχαν πραγματική δυνατότητα να εκλεγούν δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εκλογικές επιτροπές. Υπήρξε απόλυτη έλλειψη πλουραλισμού στα μέσα ενημέρωσης. Προφανώς η αντιπολίτευση είχε τη δυνατότητα να έχει χρόνο για <clears throat> πολιτικά σπότ στα μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν υπήρξε επαρκής δυνατότητα έκφρασης. Και εμείς το είχαμε επισημάνει το πρόβλημα αυτό εκείνη την εποχή. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτές οι ελλείψεις, αυτά τα προβλήματα θα μπορούσαν να επηρεάσουν και το αποτέλεσμα της εκλογικής διαδικασίας. Σε ό,τι αφορά τώρα το τμήμα της παρακολούθησης των εκλογών, ξεκινήσαμε μετά από την ε, Ολομέλεια του Στρασβούργου, όλοι μας υπογράψαμε ένα κώδικα συμπεριφοράς ως παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία μας κατά τη διάρκεια της αποστολής μας και αυτό συμπεριλαμβάνει και τη συνεργασία μας με άλλους φορείς όπως ε, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, το ΝΑΤΟ και το Οργανισμός για τη Δημοκρατία στην Ευρώπη. Αν δεν είχαμε λοιπόν κοινά συμπεράσματα με αυτούς τους φορείς, δεν θα ήταν τόσο σαφής η άποψη που διατυπώνουμε εμείς. Βλέποντας λοιπόν την κατάσταση στην Ουκρανία θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να έχει φιλοδοξίες να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό πρέπει να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν που ζητούμε, έχουμε, ζητούμε την επίτευξη ορισμένων προτύπων και από τις δικές μας χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα είναι και μία από τις χώρες οι οποίες θα ηγηθεί του ΟΑΣΕ στο μέλλον η Ουκρανία. Γι' αυτό εμείς περιμένουμε να υπάρξει μια κριτική αντιμετώπιση στην έκθεση αυτή, η οποία δημοσιεύτηκε μετά από τις εκλογές στην Ουκρανία. Δεν ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε μια τόσο επαγγελματική έκθεση και τόσο υψηλό επίπεδο και αναφέρθηκα στο θέμα αυτό και σήμερα το πρωί σε ένα άλλο χώρο. όπου ήταν παρόντες εκπρόσωποι άλλων αντιπροσωπιών παρακολούθησης. Ήμασταν στο Κίεβο, στο Νίπρο Πετρόφσκ, στο Λιεβ, την Οδυσσό και άλλες πόλεις μαζί με άλλες ε, οργανώσεις παρακολούθησης και πήγαμε και σε εκλογικά κέντρα εκτός των πόλεων αυτών. Ήταν μεγάλη η προσέλευση των εκλογέων, υψηλότερη από ό,τι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά ήταν χαμηλότερη η προσέλευση σε σχέση με το 2007, έφτανε μόνο το 62%. Υπήρξε ενδιαφέρον από την πλευρά των Ουκρανών στις εκλογές. και υπήρξε μεγάλος αριθμός παρατηρητών που ήταν παρόντες στα κέντρα, στα εκλογικά κέντρα ως διεθνείς παρατηρητές, είχαμε μια ιδιαίτερα θετικής υποδοχής. Και δεν είχαμε προβλήματα να γίνουμε αποδεκτοί ως ε, διεθνείς ε, παρατηρητές. Έρχομαι στα συμπεράσματα. Ο εκλογικός νόμος αντιμετωπίστηκε επικριτικά από πολλούς, γιατί είχε πολλές ελλείψεις που οδήγησαν σε αρνητικά αποτελέσματα. Σε ό,τι αφορά το, το διάστημα της προεκλογικής εκστατείας, υπήρξαν πολλές αρνητικές εξέλιξεις και γεγονότα. Δεν ήταν πάντα δυνατό για τους υποψηφίους <clears throat> να έχουν ισότητα συνθήκων. Και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε σε πολλά επίπεδα ήταν και το αποτέλεσμα των δικαστικών αποφάσεων που εμπόδισε σημαντικούς ηγέτες αντιπολίτευσης όπως η κυρία Τιμοσέγκο, ο Σουτσάνκο να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την ημέρα των εκλογών την ίδια, θεωρήσαμε ότι ήταν καλά διοργανωμένες οι εκλογές, δεν υπήρξαν διαταραχές της διαδικασίας της εκλογικής. Σε ό,τι αφορά την καταμέτρηση των ψήφων, στην αρχή έγινε σωστά η καταμέτρηση, αλλά σε ένα μεταγενέστερο επίπεδο δεν ήμασταν σε θέση να παρακολουθήσουμε τι ακριβώς έγινε και έχουμε πολύ σοβαρές αμφιβολίες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει, δεν έχει υπερατωθεί η εκλογική διαδικασία και επομένως δεν έχουμε τα πλήρη αποτελέσματα των εκλογών λόγω αυτού του γεγονότος σε ό,τι αφορά το τμήμα που αφορούσε την αναλογική ανάδειξη υποψηφίων, τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν ήταν πολύ κοντά στα exit polls. και τις προβλέψεις πριν από τις εκλογές, όλα αυτά ήταν συνεκτικά μεταξύ τους. Επομένως, δεν υπήρξαν καθόλου διαμαρτυρίες για το τμήμα της ε, αναλογικής εκλογής. Σε ό,τι αφορά όμως το πλειοψηφικό τμήμα των εκλογών υπήρξαν σοβαρά προβλήματα σε τουλάχιστον 12 εκλογικές περιφέρειες. Οι παρατηρητές κατα... κατέγραψαν το γεγονός ότι σε πολλές εκλογικές περιφέρειες υπήρξαν προβλήματα. Σε ορισμένε έγινε ένα αντικείμενο αγοραπολισιών η ψήφοι παρά το γεγονός ότι αυτό θεωρείται αδίκημα βάσει του ουκρανικού δικαίου. Όταν αξιολογούμε τις εκλογές αυτές θα πρέπει να θυμόμαστε ότι υπάρχει ένα σύστημα σε δύο τμήματα. Το τμήμα που είναι αναλογικό και το τμήμα που είναι πλειοψηφικό. Και αυτό επηρεάζει η μορφή αυτού του συστήματος επηρέασε και την τελική μας εκτίμηση η οποία ήταν αρνητική για την καταμέτρηση των ψήφων. Αν συγκρίνουμε την Ουκρανία με άλλα πρώην σοβιετικά κράτη, σίγουρα υποστηρίζουμε τη δυνατότητα των Ουκρανών να κάνουν τις δικές τους πολιτικές επιλογές και πράγματι ίσχυσαν το δικαίωμα επιλογής τα κόμματα της αντιπολίτευσης πήραν μια ισχυρή υποστήριξη. Αλλά μπορούμε να συγκρίνουμε αυτές τις εκλογές με τις εκλογές του 2007 στην Ουκρανία. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε προς τους Ουκρανούς σαν να, όπως αναφερόμαστε και σε ένα καλό γειτονά μας και να τους τονίσουμε ότι οι εκλογές αυτές δεν ήταν ιδιαίτερα καλύτερες από τις εκλογές του 2007 και του 2010. Και επειδή περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα, για τις εκλογές. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πράγματα δεν πήγανε ακριβώς κατ' ευχήν, όπως θα έπρεπε να είναι. Και υπάρχει και μια πρόταση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής στην Ουκρανία να επαναληφθούν για μια σειρά λόγων οι εκλογές σε πέντε εκλογικές περιφέρειες. Όλα αυτά θα μπορώ να σας τα εξηγήσω σε περισσότερο λεπτομέρεια αν κάποιος ενδιαφέρεται. Θα πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να διευκρινιστεί και να διευθετηθεί βάσει του Ουκρανικού δικαίου. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν λύσεις οι οποίες είναι νομικά <clears throat> στεγανές και στεναρές. Οποιασδήποτε αμφιβολίες πρέπει να καταλήξουν στα δικαστήρια. Επίση υπάρχουν και τα θέματα για τι μελλοντικέ αλλαγέ που θα επέρθουν στο εκλογικό δίκαιο και εκεί θα πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε όλοι τμήματα μια κοινότητα των χωρών που ανήκουν στον ΟΑΣΕ και η Ουκρανία πρέπει να τύχει αντιμετώπιση σαν χώρα με ευρωπαϊκέ φιλοδοξίε. Και φυσικά οι Ουκρανοί θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα του εκλέγην και έχουν υποστηρίξει κυρίως τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα. Σας ευχαριστώ. Πριν να, δώσω το λόγο στους αδελφούς που τον έχουν ζητήσει, να σας επιθυμίσω ότι έχει διανεμηθεί και η έκθρη. Όποιος θα θέλει να τη διαβάσει είναι στη διάθεσή σας. Ο κύριος Γκάλερ καταρχήν που ήταν αντιπρόεδρος της αντιπροσωπείας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Γκάλερ. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον ε, Παβελ Κόβαλ, τον επικεφαλής της αντιπροσωπεία μας, όχι φυσικά μονάχα για την έκθεση που μας παρουσίασε, αλλά και για την καλή ηγεσία της αντιπροσωπείας, την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι έχει συμβάλει η δική του παρουσία, ώστε να μπορέσουμε με τις άλλες τρεις, με τις τέσσερις κοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες και με τον, με τον να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια πραγματικά ουσιαστική παρακολούθηση των εκλογών και αυτό ήταν σημαντικό. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την εκλογική διαδικασία ως ένα σύνολο. Η παρουσία μας ήταν ε, μονάχα στο τελευταίο τμήμα της προεκλογικής διαδικασίας και την ημέρα των εκλογών. Μόνο αυτό το τμήμα μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε ως αυτόπτες ε, μάρτυρες και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι λειτουργήσε σωστά αυτό το τμήμα παρά το γεγονός ότι ίσως ήταν κάπως υπερβολικά γραφειοκρατικές οι διαδικασίες στα εκλογικά τμήματα. Μετά από μισή ώρα μονάχα από το τέλος των ε, της εκλογικής διαδικασίας άρχισε η καταμέτρηση, ενώ στις περισσότερες από τις χώρες μας θα είχε γίνει ήδη όλη η καταμέτρηση. Θεωρούμε όμως ότι υπήρξε μια διαφάνεια σε σχέση με την ε, ε, καταμέτρηση, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια, αλλά η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική. Τώρα αυτά τα οποία δεν μπορέσαμε να δούμε με τα δικιά μας μάτια και αυτά τα είπαν άλλοι παρατηρητές ότι υπήρξε πρόβλημα με τη μεταφορά των αποτελεσμάτων, με την ε, συνολική συγκέντρωση των αποτελεσμάτων, ενδεχομένως καταλήξαμε σε καταστάσεις όπου δεν υπήρξε ιδιαίτερη ικανοποίηση για, τα, για τον τρόπο που τον οποίο έγινε. Και ούτως ή άλλως όλη αυτή η διαδικασία κράτησε πάρα πολύ μέχρι να τροφοδοτηθούν οι υπολογιστές με τα αποτελέσματα και ώστε να χρειαστήκανε μέρες για να γίνει και η δημοσίευσή τους. Θέλω λοιπόν να επαναλάβω ότι σίγουρα μετά το τέλος της ε, σοβιετικής παρουσίας, μετά από 21 χρόνια από την αποχώρηση των Σοβιετικών, θα έπρεπε να υπάρχει μια πιο καλή εκλογική διαδικασία. Θα πρέπει να διαπιστώσουμε τις ελλείψεις οι οποίες ε, υπήρξαν στην διαδικασία αυτή. Όλα αυτά όμως δεν σημαίνουν ότι εμείς θα πρέπει να διακόψουμε τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με την Ουκρανία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο, να τον εντατικοποιήσουμε. Θα πρέπει να καταστήσουμε όμως κατά την άποψή μου κάτι σαφές, το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Δεν πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη οδό που θα σήμαινε ότι επειδή έχουμε σημαντικές ε, επικρίσεις ότι δεν θα θέλαμε να συνεργαζόμαστε πια με την Ουκρανία. Ίσα ίσα. Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε την συνεργασία με την Ουκρανία και αυτό είναι το πιο απαραίτητο. Αυτό είναι λοιπόν το δικό μου συμπέρασμα, ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, μεγαλύτερη προσπάθεια να προσελκύσουμε την Ουκρανία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα τους υποχρεώσει να τροποποιήσουν και να βελτιώσουν τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στην εκλογική διαδικασία. Δεν φαντάζομαι ότι κάποιος ο οποίος είναι σε θέση ευθύνης στην Ουκρανία θα ήθελε πράγματι να ακολουθήσει μονάχα τις επιταγές της ε, Ρωσίας. Δεν πιστεύω ότι πέραν από ορισμένου οι οποίοι ανήκουν στο φιλορωσικό κόμμα, όλη η άλλη πολιτική τάξη στην Ουκρανία θέλει να ακολουθήσει μια κατεύθυνση που υπαγορεύεται από κάποιον άλλον, από τη Μόσχα συγκεκριμένα. Πρέπει λοιπόν να τονίσουμε την ανάγκη για καλύτερα πρότυπα σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κοπήσει πάντα στα πλαίσια της ΟΑΣΕ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι θέλουμε να βοηθήσουμε την ε, Ουκρανία να κάνει τις επόμενες εκλογές με πιο επιτυχή τρόπο και σίγουρα θα θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα εφαρμοστούν πλήρως τα πρότυπα τα οποία προτείνει ο ΟΑΣΕ να μπορέσουν να εφαρμοστούν καλή την πίστη και αποτελεσματικά. Πιστεύω ότι λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε ότι για το μέλλον είναι, σημαντική να υπάρξει, είναι σημαντικό να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία με την Ουκρανία για την υποστήριξη της ε, δημοκρατίας και στα άλλα θέματα όπου έχουμε ήδη συνεργασία με την Ουκρανία, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να κινηθεί με ένα τέτοιο τρόπο, ο οποίος είναι κατάλληλος για την υποστήριξη της δημοκρατίας και όχι να υποστηρίξουμε την περαιτέρω ολιγαρχοποίηση της Ουκρανίας. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε αντίθετα την πορεία προς τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Μάλιστα, συνάδελφος Εύεριν, αλλά θα πρέπει να περιοριστείτε στα δύο λεπτά παρακαλώ οι υπόλοιποι που θα μιλήσετε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση που υπευλήθη από τον πρόεδρο της, τον επικεφαλής της αποστολής. Ήμουν και εγώ μέλος αυτής της αποστολής. Υποστηρίζω ακόμη τις δηλώσεις που έκανε επιτόπου στην Ουκρανία και το περιεχόμενο της έκθεσης το οποίο μας υπέβαλε. Συνεπώς, δεν θα μπω τώρα στις λεπτομέρειες, ούτε θα επαναλάβω τα δεδομένα της υπόθεσης. Θα ήθελα να κάνω τέσσερα πολιτικά σχόλια. Απλώς να σημειώσω ότι είναι λίγο ειρηνικό, να μιλάμε σήμερα για τα ελαττώματα της εκλογικής διαδικασίας στην Ουκρανία. Μόλις ακούσαμε ότι το Euro, ε, από το και το CNN για τα προβλήματα τα εκλογικά στη Φλόριδα. Παντού υπάρχουν προβλήματα λοιπόν. Αλλά ασχοληθούμε με την Ουκρανία εμείς. Θα κάνω σύντομα σχόλια. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται να δημιουργεί προοπτική ένταση πολιτικής στην Ουκρανία. Υπήρξαν ελαττώματα, ελλείψεις, αλλά πρέπει να αντιμετωπιστούν ορθολογιστικά, επικοδομητικά, με μια αντίδραση θετική χωρίς να γίνεται κανείς πιο ριζοσπαστικός από ότι η αντιπολίτευση και χωρίς να οδηγεί την αντιπολίτευση σε πιο ριζοσπαστική θέση. Δεύτερον, δεν πρέπει να μην χρησιμοποιήσουμε τους μηχανισμούς και τα κίνητρα τα οποία παρέχονται από τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για την εναρμόνιση της πολιτικής κουλτούρας των δύο. Είδαμε λοιπόν ότι οι πολιτικές κουλτούρες είναι κάπως διαφορετικές, αρκετά διαφορετικές. Για να μπορέσουμε, πρέπει να μπορέσουμε ταυτόχρονα να προωθήσουμε τους στόχους μας, τους γεωπολιτικούς και τους γεωστρατηγικούς. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να αποξενώνει την Ουκρανία και να την οδηγεί σε αντίθετες κατευθύνσεις από την ένταξή της στην ΕΕ. Ε, ακόμη δεν πρέπει ΕΕ να απογοητεύει τον λαό που παρά τα ελαττώματα του εκλογικού συστήματος σαφέστατα τάχθηκε υπέρ της ευρωπαϊκής ένταξης της Ουκρανίας. Χωρίς αυτή την τάση την ένταξη τίποτα σταθερό δεν μπορεί να επιτευχθεί. Ελπίζω λοιπόν ότι οτιδήποτε και αν πούμε από εδώ και πέρα πραγματικά να μην ξεχνάμε αυτές τις ανάγκες που, που πρέπει να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος Κορατσαβίλτ που ήταν ε, μέλος ε, της αποστολής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήταν ε, μεγάλη χαρά να αποτελώ μέρος της εκλογικής αντιπροσωπείας στην Ουκρανία. Θέλω να αναφερθώ στην πλήρη υποστήριξη που όλοι δώσαμε, γιατί πραγματικά ο κύριος Πάβελ ε, μας έδωσε πάρα πολλές συμβουλές, ε, ήταν ε, πολύ διαφανή η διαδικασία και όλοι θέλαμε να υποστηρίξουμε το Συμβουλίο της Ευρώπης, τον ΟΣΑΔ και το Συμβουλίο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τη δήλωση που προήλθε από όλου αυτού δηλαδή και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίσουμε ότι δεν υπήρξαν ισότιμοι κανόνε στην εκλογική διαδικασία και κυρίω είδαμε ότι υπήρξε έλλειψη ε, τη επαρκού κάλυψη από τα μέσα μαζική ενημέρωση, μειωμένη χρηματοδότηση τη προεκλογική εξτρατεία κτλ. Οι εκλογέ όμω μπόρεσαν να έχουν ε, επιλογή. Γενικά υπήρξε ηρεμία κατά τη ε, διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ε, και όπως πολύ καλά ανέφερε ο κύριος Παβέλ, ε, υπήρξε μια αξιολόγηση την επόμενη μέρα των εκλογών, αλλά εμεί τώρα το βλέπουμε ω μια εκλογική διαδικασία, όπω είπε και ο συνάδελφο δίπλα μου. Μετά τι εκλογέ είδαμε μια επιδείνωση τη κατάσταση και είδαμε ότι και η καταμέτρηση δεν μπορεί να γίνει, να ολοκληρωθεί, συνεχίζεται η διαδικασία, δεν μπορεί να αξιολογηθεί λοιπόν τόσο θετική όπως η αξιολόγηση που είχαμε την επόμενη μέρα των εκλογών. Όπως ε, είπαν ο κύριος Πέβελ και άλλοι, ε, περιγράφησαν καλά οι ελλείψεις της εκλογικής διαδικασίας, αλλά θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Νομίζω ότι είναι σημαντικό ε, να διατηρήσουμε την αξιοπιστία τη αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχήν, να συνεχίσουμε να είμαστε ενωμένοι, στο να υποστηρίξουμε μία κοινή θέση βάσει τη συνένεση. Αλλά ε, να μην ε, επιτρέψουμε καταχρήσεις ή παρερμηνίες ε, και τις θέσεις της διεθνούς κοινότητας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της αξιοπιστίας της αποστολής των παρατηρητών. Στο στάδιο αυτό είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε την εκλογική διαδικασία από τις μακρόχρονες σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι τόσο κοντά στην καρδιά μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί είναι ρευστή ακόμα η κατάσταση, έχουμε διάφορα μηνύματα, συνεχίζεται η καταμέτρηση και νομίζω ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να είμαστε απόλυτα δεσμευμένοι και να παρακολουθούμε τι σημαίνει. Ε, ο, όσα φεύγει εμεί όμω μένουμε και να μην ε, περάσουμε σε διάφορα συμπεράσματα για τι θεωρήσει, διάφορε συμφωνίε, τι σχέσει με τη Ρωσία και όλα αυτά τα στρατηγικά θέματα. Η δική μας αποστολή βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και στην αμεροληψία. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε με τη Φλόριντα, ε, ούτε να συγκρίνουμε με τη συμβαίνει στη Ρωσία και στη Λευκορωσία. Εμείς συγκρίνουμε με τα διεθνή πρότυπα των δημοκρατικών εκλογών. Και η δημοκρατία δεν είναι αλακάρτα. Ελπίζω, Πρόεδρε, να καταλήξουμε σε συνένεση σε αυτό τον Νίκο για να έχουμε μια ισχυρή θέση και μια κοινή δήλωση για την αποστολή των εκλογικών παρατηρητών. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Νάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ ήμουν μέλος της εκλογικής αποστολής και θέλω και εγώ να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την, τον κύριο Κόβαλ και να υποστηρίξω αυτά που είπε. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να προχωρήσουμε με μικρά βήματα συνεργασίας ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη προσέγγιση με την Ουκρανία, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παράθυρο ανοιχτό το οποίο θα επιτρέψει περαιτέρω θετικές κινήσεις ε, στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, γιατί το οικονομικό και πολιτικό κλίμα στην Ουκρανία δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις περαιτέρω σχέσεις μας με την Ουκρανία. Είναι σημαντικό όχι μονάχα να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ε, στην κύρωση της ε, συμφωνίας με την Ουκρανία και να υποβαθμίσουμε τις προσδοκίες μας. Θα πρέπει εμείς να δείξουμε και ισχυρή πολιτική θέληση ώστε να υπάρξουν αποτελεσματικές δομές διακυβέρνησης στην Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή η Ουκρανία δεν είναι σε θέση λοιπόν να εκπληρώσει τα υπεσχημένα σε επίπεδο καλής διακυβέρνησης. Εμείς όμως θα πρέπει να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας και εδώ πέρα το σχέδιο για τη φιλελευθερωποίηση προξενικών ε, θεωρήσεων που έχει εφαρμόσει η Ουκρανία από το 2010 είναι ιδιαίτερα θετικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι με, την, με τις προσπάθειες της Ουκρανίας μπορούμε να περατώσουμε την πρώτη φάση αυτής της συμφωνίας. Και πρέπει να ζητήσουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση των προσπαθειών. Επίσης η, Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις ε, σχέσεις με την Ουκρανία στα πλαίσια τη συμμετοχή τη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ενέργεια και επίση να χρησιμοποιήσουμε και τι ευκαιρίε αυτέ που προκύπτουν από την εταιρική σχέση. Και τέλο, θα πρέπει να υπάρξει μια πιο στενή σχέση με την κοινωνία των πολιτών τη Ουκρανίας. Και επίση για την αποστολή του Πατ Κόξ και του Κουανεύσκη σε σχέση με την ε, προσπάθεια απελευθέρωση της Τιμοσέγκο και του Λουσέγκο. Εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν θετικό να επιφορτιστεί και να, να φορτωθεί μάλλον αυτή η αποστολή αυτή με τις κατηγορίες για στρέβλωση και παραποίηση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σίεβιτς. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όσους ε, συνεχάρισαν τον επικεφαλής ε, της ε, αντιπροσωπείας μας. Πραγματικά η αποστολή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Υπήρξαν πάρα πολλά έντονα συναισθήματα γιατί είχαμε συζητήσει το θέμα της Ουκρανίας για έναν ολόκληρο χρόνο πριν τις εκλογές. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια που αναφέρθηκαν, αλλά δεν θέλω να πω ότι οι εκλογές ε, μπορούν να συγκριθούν με την κατασκευή ενός αυτοκινήτου. Μιλάμε για τεχνολογία. Η τεχνολογία των εκλογών ε, δεν ήταν πολύ καλή. Τέλεια δεν θα την ονομάζαμε. Και η προεκλογική εκστρατεία δεν ε, να από κατάλληλους κανόνες ε, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την κάλυψη των μέσων μαζικής ενημέρωσης κτλ. Αλλά οι Ουκρανοί μπορούσαν τελικά να εκλέξουν αυτούς που ήθελαν. Από τα 20 κόμματα διάλεξαν 5. Αυτό δείχνει ότι ψηφίζουν ε, με όριμο τρόπο οι Ουκρανοί και το αποτέλεσμα μας δείχνει ότι οι Ουκρανοί ήταν αποφασισμένοι να κάνουν μια επιλογή. Τώρα έχουμε ένα προϊόν. Το αποτέλεσμα αυτής της ατελούς τεχνολογίας και τα αποτελέσματα των εκλογών δεν αποτελούν ένα τέλειο προϊόν. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα προϊόν το οποίο μπορεί να λειτουργήσει. Κατά κάποιο τρόπο. Τα δύο κύρια κόμματα δεν είναι ικανοποιημένα, το κόμμα των περιφερειών δεν είναι ικανοποιημένο γιατί δεν κερδίσε την πλειοψηφία που ήθελε να κερδίσει. Η αντιπολίτευση επίσης δεν είναι ικανοποιημένη γιατί ήθελε να έχει καλύτερα ποσοστά σε σχέση με το κόμμα των περιφερειών. Η αντιπολίτευση, ακόμη και αν η ηγέτης του ήταν ε, στη φυλακή, έδωσε μεγάλη μάχη οι εκλογές ουσιαστικά ήταν ε, ένα είδος δημοψηφίσματος για την ε, φυλάκιση, σχετικά με τη φυλάκιση της Γιούλια Τιμοτσένκο. Σας παρακαλώ. Θα ήθελα να μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμα, 30-40 δευτερόλεπτα. Τελειώνω, Πρόεδρε, τελειώνω. Επομένως, είχαμε δύο νέα κόμματα που μπήκαν στο Κοινοβούλιο. Το κόμμα του κυρίου Κλίτσκο, που είναι φιλοευρωπαϊκό, μπήκε στο κοινοβουλίο, πολύ θετικό, και το Σβομπόντε, το οποίο είναι ξενοφοβικό, εθνικιστικό κόμμα. Και η παρουσία του στο κοινοβούλιο θα οδηγήσει σε προβλήματα. Η ερώτηση λοιπόν είναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αγοράσει αυτό το προϊόν, τα αποτελέσματα των εκλογών, με όλες τις ελλείψεις που παρουσιάζει και τα μειονεκτήματα είδαμε ότι πρέπει να επαναληφθούν οι εκλογές ε, σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Ο κύριος ε, Τάνοκ, ε, σας παρακαλώ να είστε πολύ συνοπτικός. Θα είμαι σύντομο πρόεδρε. Βεβαίω υποστηρίζω την έκθεση. Με ενδιαφέρει το σχόλιο ότι 58% είναι μεγάλη συμμετοχή. Αυτό θα ήταν πολύ το χαμηλότερο ρεκόρ για την χώρα μου. Συνεπώς είναι ενδιαφέρον πως υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις ως προς τη συμμετοχή. Βεβαίως η υπόθεση Τιμοσέγκο δεν βοηθά στο να προχωρήσουμε με την υλοποίηση της σχέσης ε, της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης και η ρεγιόν, το κόμμα των περιφερειών δηλαδή έχει μόνο 223 έδρες Τώρα, ακόμη και αν εξαγοράσουν ε, όποιον μπορούν και θέλει, ε, δεν μπορούν να φτάσουν στους 300 που απαιτούνται για πλειοψηφία. Αυτό συνεπώς είναι ένα μήνυμα προς την αντιπολίτευση που έχει 50% και κάτι ακόμη από την ψήφο του λαού. Ε, θα αμφισβητήσουν λοιπόν την κυβέρνηση Ανικόβιτς η ερώτησή μου προς τον Πάβελ αφορά τις 12 έδρες που πιθανόν, για τις οποίες πιθανόν να επαναληφθεί η εκλογή. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να στείλουμε και μια άλλη αποστολή και ειλικρινά λυπάμαι ότι δεν, που δεν ήμουνα μαζί σας. Έχω πάει στην Ουκρανία, από τότε που ε, ε, έγινε η πρώτη επανάσταση ε, αλλά μπορεί να έρθω μαζί σας για να μπορέσω να διαπιστώσω τη δημοκρατικότητα. Ευχαριστώ. Συνάδελφοι, δυστυχώς έχουμε καθυστερήσει και πρέπει να αποχωρήσουν οι διερμηνείς. Μπορούμε να συνεχίσουμε μεταξύ μας τη συζήτηση αν θέλετε. Ευχάριστο θα είναι, αλλά έχει πολύ αποτελεσματικό. Θέλει ο κύριος Γκάλερ να πει κάτι. Είναι πολύ επιτακτικό, τόσο μεγάλη ανάγκη. Μάλιστα, δεν χρειάζομαι καν τους διερμηνείς, λέει ο μιλητής. Δεν ε, θα δεκτώ μια συνδηλώση από τον κύριο Σιβίτσε που κάνατε και πριν τις εκλογές ε, στην παρουσία του, παρουσία του ΕΛΜΑ και αυτός μόλις είχε τη τότε και ε, είχατε πει ότι ότι δεν, έχει, δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι είναι στη φυλακή η επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Όχι, δεν έχετε δίκιο. Δεν ήταν ελεύθερες οι εκλογές γιατί δεν μπορούσαν όλοι να συμμετέχουν ε, και δεν θα ήθελα ε, να υπάρξει τέλος πάντων ε, μια τέτοια υπόνοια για το αν ο επικεφαλής, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή. Δεν έχει κανένα νόημα. Θα ήθελα να σας καλέσω όλους να πιούμε ένα ποτό όλοι μαζί, λέει ο Πρόεδρος. Παρακαλώ, μπορείτε να πείτε την άποψή σα, αγαπητέ συνάδελφε. Αλλά ένα λεπτό, να έχετε υπομονή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στο συνάδελφο που έχει δει στο κατάλογο το λόγο και μετά θα επανέλθω σε εσά. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Κόβαλ για το έργο του ως επικεφαλής ε, της αντιπροσωπείας. Ε, μέχρι σήμερα δεν είναι σαφής η κατάσταση στην Ουκρανία γιατί η αντιπολίτευση ε, στην αρχή ήταν ε, κατά της αναγνώρισης των εκλογικών αποτελεσμάτων κατόπιν άλλαξε γνώμη το βράδυ και νομίζω ότι πρέπει να συγχαρούμε τον Μπάβελ. και αυτό είναι το πρακτικό μου αίτημα, να έχουμε μια ειδική συνάντηση ε, είτε η Επιτροπή είτε το διευρυμένο Προεδρείο με τους ε, Κόβαλ και Φασέλσκι μετά από την ε, τρέχουσα αποστολή στην Ουκρανία για να αναλύσουμε την πολιτική κατάσταση. Μάλιστα, μπορείτε να έχετε μία ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό με τον κύριο Μπρόκ, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Σιβιεβίτς. Για να... να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Γκάλερ. Εγώ δεν επιμένω, απλώ περιγράφω μια κατάσταση παρά το γεγονός ότι οι ηγέτε της αντιπολίτευσης ήταν στη φυλακή, η αντιπολίτευση είχε αρκετή δύναμη να συμμετάσχει στι εκλογές και να πετύχει ένα καλό αποτέλεσμα για την Ιουλία Τιμοσέγκο. Εμείς διαμαρτυρηθήκαμε με ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου πέρσι. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα για το πώς εμείς αντιμετωπίσουμε το θέμα της φυλάκισής της. Παρ' όλα αυτά, η κυρία Τιμοσέγκο χρησιμοποιήθηκε ως προμετωπίδα κατά κάποιο τρόπο στην εκστρατεία της αντιπολίτευσης. Επομένως, απλώς σας περιγράφω την κατάσταση ως είχε. Thank you, colleague. With your... Ευχαριστώ, αγαπητέ συνάδελφε. Σας ζητώ να μου επιτρέψετε να αποχωρήσω, λέει ο Πρόεδρος.